Buenas tardes. Καλό σας απόγευμα. Si les parece, comenzamos. Να ξεκινήσουμε αν συμφωνείτε. Entre otras cosas porque luego siempre empezamos. Γιατί πάντοτε έργουμε να ξεκινήσουμε και μετά πρέπει να τρέχουμε. A ver, por favor, un poco de silencio. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Yeah, Bueno, bueno, ahora sí, vamos. Es quiet, please. Vamos a comenzar. Να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, αν συμφωνείτε. να δούμε την ημερησία διάταξη της Επιτροπής μας, αλλά αν μου επιτρέπετε να πω ότι πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση σήμερα και είναι μεγάλη χαρά η δική μου αλλά και όλων ε, των μελών της Επιτροπής μας, γιατί θα έρθει ο κύριος Βαλέσα, ήρθε ο κύριος Βαλέσα μετά από το σοβαρό ατύχημα που είχε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ και αν ε, μου επιτρέπετε θα σας διηγηθώ και μια ειστηρία γιατί το συνάντησα σήμερα το πρωί στο Σανσέρ και δεν το φανταζόμουν ότι ήδη είχε επιστρέψει εδώ και μάλιστα όπως ε, ήλθε και το γνώρισα χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι είχε επιστρέψει ο κύριος Βαλεσό και ήταν σημαντικό λάθος δικό μου αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μεταξύ μας. Πραγματικά καλώς ήρθατε. Λοιπόν, για να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ. E, e, Ευχαριστώ. Θερμά όλους τους ε, συναδέλφους. Ευχαριστώ την κυρία Φράγα, την κυρία Βενέρα. Πραγματικά, ε, όταν ακόμη ήμουνα στο νοσοκομείο, με ενθάρρυναν ε, με τα ζεστά τους λόγια, με υποδέχτηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο. Ανυπομονώ να επανέλθω στις εργασίες της Επιτροπής μας. Μάλιστα, έτσι θα γίνει. Πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Ε, Έχουμε μία σειρά αλλαγών στην ημερησία διάταξη που έχουν τεθεί σε σχέση με τα σημεία 15, 16 και 17 που θα τα δούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Απριλίου, αν συμφωνείτε. Αυτό μας γνωστοποίησαν. Έτσι λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τα θέματα στην επόμενη επιτροπή. Λοιπόν, για να εγκρίνουμε τα παρακτικά, 27-29 Φεβρουαρίου 2012 εγκρίνονται αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας. ανακοινώσει του Προέδρου δεν έχω. Κάποια ανακοίνωση πέρα από τα όσα γνωρίζετε ήδη. Και να περάσουμε επομένω κατευθείαν στο σημείο 4, τροποποίηση του κανονισμού 1300-2008 για τη θέσπιση πολιτικού σχεδίου, για το απόθεμα Ρέγκα που κατανέμεται δυτικά τη Σκωτία και για την αλία αυτού του αποθέματο. Όπω γνωρίζετε, ήδη η Κομισιόν στι 25 ε, Ιανουαρίου μα παρουσίασε την νομοθετική πρόταση. Το Φεβρουάριο είχαμε μία σύντομη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και σήμερα ο εισηγητή θα μα παρουσιάσει το σχέδιο της ε, γνωμοδότησης και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 26 Μαρτίου το μεσημέρι. Αυτή είναι λοιπόν η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Κύριε Στίβενσον. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο στόχος της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρε, είναι ο κείμενος κανονισμός να ευθυγραμμιστεί με το νέο πλαίσιο Επίση, ε, έδραξαν την ευκαιρία για να προτείνουν και κάποιες ε, βασικές ε, τροποποίησει στον κείμενο του κανονισμού. 14 το αριθμό που συνάδουν με τα όσα υπόθηκαν εδώ στην Επιτροπή μας στην προηγούμενη συνεδρίαση το Φεβρουάριο. Σε σχέση τώρα με τη γεωγραφική τοποθεσία του αποθέματος, η τροπολογία 9 διατηρεί την τωρινή διατύπωση, ούτω ώστε σαφέστατα να προσδιορίσουμε αυτή την περιοχή ε, όπου είναι εφαρμοστέο αυτό το ε, πρόγραμμα. Ε, Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνεί σχετικά με τα οστρακοειδή ε, ε, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μην ανησυχείτε, λέω στρεφόμενος προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε ρυθμίσει όλα αυτά που είχαμε πει. Ε, κατόπιν, ε, μείωση του ποσοστού θνησιμότητας με τη βάση υπολογισμών που γίνονται με την βιομάζα, το άρθρο 7 δηλαδή, ε, δυστυχώς δεν αναφέρονται τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασίζονται. Αντίθετα, η τροπολογία 10 επανεισάγει τη διατύπωση του κείμενου κανονισμού ότι ε, οι επιστημονικές ε, συμβουλές πρέπει να προέρχονται από επιστήμονες και εγώ προσέθεσα ε, σε πλήρη διαβούλευση με τον Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Οργανισμό για τα πελαγικά είδη, γιατί από εκεί προέρχονταν τα στοιχεία. Αυτό το, αυτός ο πελαγικός λοιπόν, περιφερειακός οργανισμός έκανε τις προτάσεις ε, για τη Ρέγκα στην, ε, στα δυτικά της Σκοτίας επειδή παραμένουν τα τωρινά επίπεδα ε, και προβλέπονται πλέον πράξεις κατ' εξουσιοδότηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ώστε να δράει χωρίς καμία καθυστέρηση τελευταία. Συμφωνούμε επίσης με αυτά που είπατε για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και την αιτήσια διαβούλευση να την καταργήσουμε. Αντίθετα να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια αναθεώρηση. Ούτως ή άλλως αυτό προβλεπόταν ετησίως ένα ζητούνται συμβουλές δεν εφαρμόστηκε ποτέ και βάσει τη συνήθω νομοθετική διαδικασία ενδείκνυται να έχουμε μια τετραετή περίοδο αναθεώρηση. Επανησύγατε και τον διάταξη του κείμενου κανονισμού ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά συμβουλές από το ε, Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Οργανισμό για τα πελαγικά, γιατί αυτό προβλέπεται στη διαδικασία, καθώ και από τα επιστημονικά συμβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Στίβενσον. Με το σχέδιο εκθεσή σα, ε, με πολύ ακρίβεια μα παρουσιάσετε την προβληματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τα πολιετή σχεδία είναι τη Κομισιόν και του Συμβουλίου, αλλά και το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα γνωμοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν στα πολιετή σχέδια προσαρμόζονται τα σχέδια εγχείρησης. και συμφωνήσαμε η Κομισιόν να μπορεί να έχει την αρμοδιότητα να παρουσιάσει κατεξιοδότηση πράξης, ε, αλλά το σημαντικό είναι να μπορεί και το Κοινοβούλιο να αντιδράσει και αυτό το κάνουμε πρώτη φορά με το πολιετές σχέδιο για τη Ρέγκα. που κατανέμεται στα δυτικά της Σκοτίας. Αυτό που μας είπε ο κύριος Στίβενσον είναι πολύ σημαντικό ότι ο γεωγραφικός ε, καθορισμός, ε, και που βρίσκεται δηλαδή αυτός ο πληθυσμός, αυτό το απόθεμα, αυτό πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, με αριθμητικά στοιχεία. Σίγουρα μπορούμε να το προσδιορίσουμε και με GPS στοιχεία, αλλά πρέπει να είναι σαφές το, το για πράγμα μιλάμε. Σε αυτά τα αποθέματα πρέπει να καθορίσουμε το σημείο που βρίσκεται το απόθεμα αυτό και σιγά σιγά πρέπει να διορθώνουμε. Τα λάθη του πρέπει να έχουμε στοιχεία για όλα τα αποθέματα και τα αποθέματα που αφορούν τα πολυετή προγράμματα διαχείρισης και συγκεκριμένα για το απόθεμα της Ρέγκα στα δυτικά της Σκοτίας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό να είναι τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΡΑΚ των πελογικών ειδών που θα συμμετέχει στη διαβούλευση. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να γίνεται μια εξέταση και να παρουσιάζονται στοιχεία κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτό μπορούμε να το δεκτούμε. Και σε γενικές γραμμές αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει καμία δυσκολία να εγκριθεί με ευρία πλειοψηφία η έκθεση αυτή. Κυρία Λεβάν. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλα αυτά που έκανε. Είναι όντως ε, πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για όλα τα μελλοντικά ε, προγράμματα διαχείρισης ε, και την ευθυγράμμιση με το περιεχόμενο της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, υπάρχει μία ουσιαστική αλλαγή που έκανε ο εισηγητής. Ε, δηλαδή η γνωμοδότηση των ΣΤΕΚΦΕ και των σε αυτών των περιφερειακών γνωμοδοτικών οργανισμών. Είχε προτείνει η Επιτροπή ότι όταν δείχνουν ε, τα επιστημονικά δεδομένα πως ε, παρά είναι υψηλή η θνησιμότητα των ψαριών, προβλέπεται αυτή η αλλαγή και προτείνει ο εισηγητής το ΣΤΕΚΦΕ, το Επιστημονικό Συμβούλιο δηλαδή, να εκδίδει την γνωμοδότηση αυτή. Κατόπιν ευρεία διαβούλευση με ε, τους αρμόδιους γνωμοδοτικούς οργανισμούς. Ε, δεν έχω καταλάβει τι εννοεί όταν λέει ευρύτατη διαβούλευση με τα ΡΑΚΣ, με τους περιφερειακούς γνωμοδοτικούς οργανισμούς. Είναι προφανές ότι οι οργανισμοί πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ούτως ή άλλως το γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση προτού καν αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πράξη όμως τι σημαίνει αν έχουμε αυτή τη διατύπωση μέσα σε, σε ένα νομοθέτημα που θα λέει ότι προβλέπεται ε, ευρία πλήρης διαβούλευση, full consultation λέει στα αγγλικά. Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω τι εννοεί ο εισηγητής. Αυτή η έμφαση που δίνουμε στο ΣΤΕΑΚ που είναι επιστημονική, τεχνική και οικονομική ε, επιτροπή η οποία αξιολογεί τα αποθέματα από διαφορετικές ε, οπτικές γωνίες και παίρνει διαφόρων ειδών δεδομένα υπόψη. Όταν, παραδείγματος χάρη, εξετάζουμε αμυγός την ε, βιολογική κατάσταση του αποθέματος, ε, υποθέτω ότι στα στατιστικά δεδομένα για την εθνισιμότητα των ψαριών είναι και τα πλέον κατάλληλα δεδομένα που πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τα δεδομένα και γνωμοδοτήσεις ε, της Επιστημονικής, Κοινωνικής και Τεχνικής Επιτροπής ή των περιφερειακών γνωμοδοτικών των οργανισμών αυτά, αλλά πιστεύω ότι πάνω κάτω συμφωνούμε όλοι με τη γραμμή του εισηγητή. Ο κ. ο κύριος Καντέλα από την Κομισιόν. Καντέλα, perdón. Η κυρία Καντέλα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς ε, ήθελα να επενθυμίσω ότι εξηγήσαμε για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι αλλαγές και όπως προκύπτει από τις παρεμβάσεις φαίνεται να πηγαίνουν πιο μακριά από την απλή ευθυγράμμιση του κειμένου με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Απλώς να επαναλάβω ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση από την πλευρά της Κομισιόν να αλλάξει το ουσιαστικό περιεχόμενο του κειμένου. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να πούμε, όπως το έκανε ο εισηγητής, ότι σε ό,τι αφορά την περιοχή είμαστε απόλυτα ευέλικτοι σε ό,τι αφορά τώρα τις προηγούμενες διαβουλεύσεις, στην πραγματικότητα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ότι αυτό που προσπαθήθηκε με τις τροπολογίες ήταν να υπάρχει ώστε να δω περισσότερη ευθυγράμμιση για τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των οργάνων για τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση που έχουμε καταξουσιοδότηση πράξης. Ε, να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο πρότυπο εκτιμώντας που προβλέπετε και στη δική μας πρόταση, το υπαριθμόν 5 και θα σας το διαβάσω στα αγγλικά και λέει είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να κάνει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προσκευαστικού του έργου και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Πρόκειται για μια διατύπωση η οποία εξηγεί ότι καθώς είναι πρότυπο το κείμενο που καλύπτει όλες τις πολιτικές και καθώς αυτό είναι ένα εγχείρημα που πηγαίνει πολύ πιο πέρα από την πολιτική αλίας αλλά καλύπτει και άλλες πολιτικές ε, και ε, όλα τα τμήματα ακολούθησαν το ίδιο μοντέλο πάνω κάτω. Μιλάμε για κάτι πολύ ευρύ. Είναι προφανές ότι η Κομισιόν στο πλαίσιο αυτό που βρισκόμαστε και διαβουλεύεται και το επιστημονικό και το επιστημονικό τεχνικό και οικονομικό συμβούλιο και καταρχήν έχουμε μία ε, τεχνική διαβούλευση και κατόπιν υπάρχει μία αξιολόγηση ομοτήμων από το STCF. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντίρρηση από την πλευρά της Κομισιόν για τις διαδικασίες η αντίδραση είναι κάπως διευρυμένη γιατί πρόκειται για οριζόντιο εγχείρημα στην Κομισιόν και δεν περιορίζεται στον τομέα της αλίας. Όμως εγώ νομίζω ότι είναι δυνατό να πούμε ότι η Κομισιόν πραγματικά δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα θέματα που έχουν αναφερθεί σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και θα περιμένουμε να δούμε πώς, τι μορφή θα πάρουν οι τροπολογίες που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο και τότε θα αντιδράσουμε επισήμω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Στίβενσον. Thank you very much and thank... Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές καθώς και την κυρία Καντέλα για τις παρατηρήσεις τους σε σχέση με αυτό που μας είπε η Ζαμπέλα. Το μόνο που λέω και νομίζω ότι ε, το εξήγησε πολύ καλά τη διαδικασία η κυρία Καντέλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, λεγόταν στην αρχή ότι προβλέπεται αιτήσια αναθεώρηση στο παρελθόν, όμως ποτέ δεν συνέβη αυτό. Και λέω λοιπόν, συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τετραετία αναθεώρηση, αλλά σε μπλακούν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί. Ας ε, λάβουμε υπόψη τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Οργανισμού ε, για τα πελαγικά είδη. προσθέσουμε αυτό στην ε, αναθεώρηση που θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και όπως είπε η κυρία Καντέλα, ούτως ή άλλως ε, θα γίνεται και αξιολόγηση από ε, τους ομοτήμους αλλά και από το ΣΤΕΦΚΑ, αυτή την Επιστημονική, Κοινωνική και Τεχνική Επιτροπή. Όλα θα λαμβάνονται υπόψη. Ο κύριος Κουνή είπε στην παρέμβασή του πολύ σωστά ότι το ότι συμφωνούμε να ε, δώσουμε την αρμοδιότητα για πράξη κατά εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρα πολύ σημαντικέ επιπτώσεις για τα λοιπά πολιετή ε, προγράμματα διαχείρισης που μας απασχολούν και για το σκουμπρί ε, όλο ιδιαίτερο που έχει γίνει ένας ιερό πόλεμος ουσιαστικά στι διαπραγματεύσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη κάτι και την ε, Ισλανδία. Νομίζω πάντω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση. Λοιπόν, προθεσμία για τι τροπολογίε 26 Μαρτίου, το υπενθυμίζω. Πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, ε, το σημείο 5. Ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της κοινή ελεκτική ε, πολιτικής και είχαμε δύο φορές ανταλλαγή απόψεων το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο και την παρουσίαση ενός εγγράφου εργασία που, ανέλαβε, που έχει αναλάβει συγγήτρια τον Ιανουάριο. Τώρα η κυρία Λοβέν θα μας παρουσιάσει το σχέδιο της γνωμοδότησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, τελικά έχουμε το σχέδιο της έκθεσης ε, έτοιμο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα σας τα πω διεξοδικά. Καταρχήν, Θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ως μια μεγάλη ελευτική δύναμη εκτός των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ως ε, τη, μια πολύ μεγάλη αγορά εισαγωγής ως ε, τη μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών στον κόσμο και αυτό θέτει πολύ μεγάλη ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει ότι ε, είναι οικολογικό το αποτύπωμά τη στην αλία είτε εμείς ίδιοι τα αλλιεύουμε τα ψάρια είτε τα καταναλώνουμε μέσω αγωγών. Θέλουμε στη συνέχεια να καλωσορίσουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν και πιστεύουμε ότι οι προτάσεις σε αυτή την ανακοίνωση είναι πάρα πολύ θετικές. Πράγματι τονίζεται η ευθύνη του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκτός των δικών μας υδάτων, αλλά θεωρούμε ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι επαρκώς ευρύ, και έτσι λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και σε άλλα θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση, όπως οι εισαγωγές ε, και οι ιδιωτικές συμφωνίες, οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, από τις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από όσους αλλιεύουν υπό άλλες σημαίες. Βασικά πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ή εκτός ε, των υδάτων της Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται στα ίδια πρότυπα σε ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονομική αηφορία και τη διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, οι ίδιοι κανόνε θα πρέπει να ισχύουν ε, για τι επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αλλιεύουν εντό είτε εκτό των υδάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θεωρούμε ότι οι στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής διάστασης της κοινή ελευθερικής πολιτικής θα πρέπει να αναφερόνται στο βασικό κανονισμό, δηλαδή στο νομικό κείμενο. Ε, τώρα είναι πάρα πολύ μινιμαλιστικό το κείμενο αυτό και χαίρομαι να πω που χθε το Συμβούλιο συμφώνησε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εξωτερική πολιτική συμφώνησαν ότι οι βασικοί στόχοι και οι αρχές της ε, εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αναγράφονται στο βασικό κανονισμό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα καταθέσουμε προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση στο μέλλον στην έκθεση Ρόντουστ. Οι γενικές ε, διατάξεις ε, σχετικά με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως. Τώρα, από, τα σημεία 5 το σημείο, το σημείο 5 στο σημείο 10, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι δράση πρέπει να αναλάβει σε επίπεδο ΙΕ και επίσης αναφερόμαστε στην καταπολέμηση της ε, αλίας ε, πλά, της, αλίας, ε, της παράνομης λαθρής και ανέρχης αλίας παγκοσμίω και πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με κύριους εταίρους όπως η Ιαπωνία, η Πακεκίνα. Επίσης πιστεύουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν στην ανακοινώσή της ε, να δημιουργήσει ε, ένα καθολικό σύστημα τεκμηρίωσης για τα ελεύματα είναι καλό. Το Συμβούλιο δεν το αναφέρει αυτό στο Συμβούλιο, Συμβουλίου, αλλά εμείς ε, θέλουμε να εγκρίνουμε αυτή τη φιλοδοξία της Κομισιόν και επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο ενεργή σε επίπεδο ΟΗΕ για να διερευνήσει μέσα έτσι ώστε η παγκόσμια κοινότητα να συστήσει ε, καλύτερη διακυβέρνηση των, και συστήματα διακυβέρνηση των ωκεανών που να καλύπτουν και τους θαλάσσιους πόρους αλλά και άλλους πόρους που, αυξανο, που εκμεταλλευόμαστε το ένα και περισσότερο. Έρθουμε τώρα στις διμερείς ελευτικές συμφωνίες. Η Κομισιόν της αποκαλεί βιώσιμες ε, Αλευτικές συμφωνίες την ανακοίνωση και το Συμβούλιο διατήρησε το όνομα Fisheries Partnership Agreements στα συμπεράσματα, δηλαδή αλευτικές συμπράξεις. Ε, εδώ εμείς δεν έχουμε ονοματίσει, δηλαδή υπάρχουν ε, διαφορετικοί όροι που περιγράφονται, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η συμφωνία ε, ωφελούν ε, και τα δύο μέρη, δηλαδή ε, όχι μόνο το παράκτιο κράτος. Αλλά φυσικά σε κάποιο βαθμό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτή τη συνεισφορά ε, των ψηλιών ως ε, εφοδιασμό στα τρόφιμα, αλλά δεν νομίζω ότι εισάγουμε πάνω από το 60% των ψαριών. Έτσι λοιπόν ε, δεν συνεισφέρουμε στην επιστημιστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις χώρες εταίρου με τι οποίε έχουμε ελευτικέ συμφωνίε. Και επίσης ε, είναι σημαντικό να παρέχουμε υποστήριξη στον κλάδο για την εποπτεία, της ε, επιστημονικής αξιολογήσεις και επίσης για την οικοδόμηση υποδομών στις χώρες αυτές. Βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι ε, παλιές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, δεν ε, έχουν ε, προποθέσει. προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις λοιπόν και έχουμε κάποιες βασικές αρχές. Μία είναι ότι πρέπει να υπάρχει πλεόνασμα τσαριών στα ύδατα του παράκτου κράτους, που το ίδιο δεν έχει την ικανότητα να αλλιεύσει και δεν το χρειάζεται το απόθεμα αυτό για τη δική τους επιστημιστική ασφάλεια. Και όταν έχει αποδεικτεί αυτό αποτελεσματικά, επιστημονικά, μόνο μπορεί να διαπραγματευτεί, μόνο τότε μπορεί να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση σε αυτά τα ύδατα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι το κράτος με τον οποίο πραγματευόμαστε τις αλλιευτικέ ευκαιρίε ε, πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές. Αλλά πρέπει να υπάρχει ε, στις ε, συμπράξει αυτές και μία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, πιστεύουμε ότι η ρήτρα πέρι αποκλειστικότητα είναι πολύ σημαντική, πρέπει να διατηρηθεί όταν ε, έχουμε μία λευτική συμφωνία με μία τρίτη χώρα, δεν θα πρέπει να, είναι, να υπάρχουν ε, ιδιωτικές συμφωνίες με τις επιχειρήσεις. Όλοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της αληφτικής συμφωνίας. Και επίσης ε, στην ανακοίνωση της Κομισιόν τονίζεται το θέμα της ε, κατάχρησης της αλλαγής σημαίας, ε, flag hopping, όταν ε, οι επιχειρήσεις της Ένωσης αλλιεύουν δυνάμεις συμφωνιών που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν αλλάζουν σημαία, πάνε σε ένα άλλο κράτος και συνεχίζουν να αλλιεύουν στα ύδατα κίνηση της χώρας ή κάπου αλλού και μπορούν να επανέλθουν στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουν να αλλιεύουν δυνάμει της Ελευτικής Συμφωνίας ή δυνάμει πλαισίου πόδα. Αυτό αποτελεί πρόβλημα γιατί εμείς θέλουμε να ελέγχουμε τόνους, ε, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ίδια ευθύνη για την αηφορία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι πρέπει να υπάρχει πλεόνασμα δηλαδή του πληθυσμού, των ψηλίων κτλ. Και δεν θα πρέπει να κρύβονται πίσω από διαφορετικές σημαίες. Έτσι λοιπόν αυτό που προτείνουμε είναι ο κανονισμός για την ελευτική άδεια να τροποποιηθεί έτσι ώστε ε, τα σκάφη που έχουν σημαίνει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωρινά έχουν εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσουν ευκαιρίε αλλού να μην μπορούν να υποφεληθούν ε, τέτοιων ευκαιριών δυνάμει ε, των ελευτικών συμφωνίων αν θέλουν να επανέλθουν στο μητρό, στο μυολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αυτού. Και θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία των ε, συνθήκων εργασίας ε, πρέπει να συμπεριλάβουμε εκεί και το σεβασμό του σύσταση 188 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας και τις συστάσεις του ΕΛΟ. Επίσης, χρειαζόμαστε διαφάνεια για την συνολική απόσυρση των ε, ψαριών στα ύδατα της τρίτης χώρας. Πρέπει να ξέρουμε ποιος άλλος αλλιεύει εκεί, πόσα ψάρια αλλιεύονται και από το τοπικό στόλο ή από άλλες χώρες, είτε μιλάμε για ιδιώτες είτε για άλλες χώρες. Και φυσικά τα σκάφη της Ένωσης δεν θα πρέπει ποτέ να ανταγωνίζονται για να λιεύουν τους ίδιους πόρους με τον τοπικό στόλο. Αυτό δεν είναι καθόλου αποδεκτό. Για να επανέλθω στο θέμα του πλεονάσματος, ένα από τα προβλήματα για να δημιουργηθεί το πλεόνασμα, μάλλον να δούμε αν υπάρχει πλεόνασμα, είναι ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα βέβαια. Αν δεν ξέρουμε πόσα ψάρια αλλιεύονται συνολικά από όλου του τόλου, δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοια δεδομένα αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους σπόρους ε, για τους επιστήμονες. Και πιστεύουμε ότι θα ήταν ε, καλό ε, να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια ερευνητικά σκάφη σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο στόλος και να διερευνήσει τα θέματα αυτά που αποτελούν ε, προπόθεση για οποιαδήποτε ελευτική συμφωνία. Ένα άλλο σημείο που στηρίζουμε την πρόταση τη Κομισιόν και το Συμβούλιο ήταν θετικό επίση χθε ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι η αποσύνδεση των πληρωμών. Δηλαδή έχουμε μία ενίσχυση, μία πληρωμή για που αφορά την ε, πραγματική πρόσβαση στους πόρους και έχουμε και άλλη μία πληρωμή που αφορά την ε, τομεακή υποστήριξη. Και πιστεύουμε ότι η πληρωμή για την πρόσβαση θα πρέπει να καταβάλλεται από τους ίδιους τους πλειοκτήτες, θα πρέπει να πληρώνουν ε, ένα δίκαιο μερίδιο βάση και τον τιμό της αγοράς για την πρόσβαση του στόλου μάλλον για τα τέλη πρόσβασης, με συγχωρείτε, και για το θέμα της διαφάνειας, ε, το Κοινοβούλιο η Κοινωνία των Πολιτών, όλοι θα πρέπει να ενημερώνονται πολύ περισσότερο επί των όρων των συμφωνιών. Θέλουμε οι αιτήσει εκθέσεις να στέλνονται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο Θέλουμε επίσης το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην διαδικασία της διαπραγματεύσης και να παρακολουθεί την θέση σε λειτουργία των συμφωνιών και πιστεύουμε ότι οι συνεδριάσεις των μεικτών επιτροπών θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκπροσωπείται εκεί. Θα πρέπει να εκπροσωπείται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξέρουμε ότι η διαφάνεια είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Και μόνο αν θέσουμε το παράδειγμα ότι είμαστε απόλυτα διαφανείς σε σχέση με την ε, λήψη των πόρων και τις πληρωμές και την παρακολούθηση της ε, τομέας ενίσχυσης, ε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταλήξουν τα χρήματα στις τσέπες κάποιων και η κοινωνία των πολιτών στις τρίτες χώρες να ενημερώνεται πλήρως για το τι συμβαίνει, για το ποιος ε, αλλιεύει, πόσα σκάφη, τι πιάνουν και πόσα πληρώνουν. Επίσης, πιστεύουμε ότι μια περιφερειακή προσέγγιση στην διαπραγμάτευση των λευτικών συμφωνιών είναι μια καλή ιδέα, καθώς ε, τα ψάρια μετακινούνται ε, μεταξύ των εθνικών συνόρων και ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε την περιφερειοποίηση της ε, διαχείρισης ε, των αποθεμάτων και ορισμένε από τις χώρες στη Δυτική Αφρική, λόγου χάρη, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών, αλλά τα αποθέματα των ψαριών μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν αγοράζουμε ένα πλεόνασμα δύο ή τρει φορές που τη μία φορά είναι στη Μαυριτανία, την άλλη στην Γουινέα και στη Σενεγάλη, κατόπιν με την οποία δεν έχουμε συμφωνία βέβαια. Αυτά για τι αλευτικέ συμφωνίες. Να περάσουμε τώρα στη Σπόδα. Ασχολήθηκα επί μακρόν με αυτό το θέμα μέσα στην έκθεση για την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλλά είναι ιδιαίτερα ε, ε, σημαντικοί αυτοί οι οργανισμοί, διότι διαχειρίζονται τα άκρος μεταναστευτικά ήδη. Μιλάμε για ψάρια πώς επιτοπλίστων πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη και μένουν σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πρόκειται για διεθνείς ε, πόρους και οφείλουμε να τους διαχειριζόμαστε με σοβαρότητα. Αυτή η περιφερειακή οργανισμή διαχείρισης ε, αλίας είναι τα μόνα φορά, τα μόνα οι μόνοι οργανισμοί που υπάρχουν ε, που δύναται να διαχειριστούν ε, αυτό το κοινό για ολόκληρη την ανθρωπότητα κληροδότημα. Πρέπει να προφυλάξουμε τα αποθέματα για τις επόμενες ε, γενιές και να εξασφαλίσουμε μια ίση δίκαιη κατανομή των αποθεμάτων ανάμεσα στις στοχές και τις πλώσιες χώρες, ανάμεσα στα παράκτια κράτη και όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ καλή διαπραγματευτική θέση για να προσπαθήσει να ενισχύσει ε, τις αρμοδιότητες ε, των πόδα. και είναι και μέλος ε, στους πιο σημαντικούς πόδα, οπότε μπορεί να ενισχύσει τη δράση τους. Κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να μεριμνήσουμε ώστε να τακτικά ανεξάρτητοι οργανισμοί να αναθεωρούν τα καταστατικά των πόδα, να βελτιώνεται το σύστημα λήψης αποφάσεων. Επίσης, διεύρυνση της κάλυψης πρέπει να επιδιώξουμε, ώστε να διαχειριζόμαστε όλα τα ε, αποθέματα βάσει μιας οικοσυστημικής προσέγγιση. Ο εύξηνο πόντο επίσης θα υποφεληθεί πάρα πολύ από τη σύσταση ενό νέου περιφερειακού οργανισμού. Το θέμα της ε, κατανομής στο εσωτερικό των ΕΠΟΔΑ είναι επίσης ένα θέμα που θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Έχουμε τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες που πραγματικά διεκδικούν ε, το μερίδιό τους από αυτά τα διεθνή ηχθή αποθέματα και ε, τα ιστορικά μέτρα αναφορά για τον υπολογισμό των αλλιευμάτων γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ο μόνος συντελεστής ε, στον υπολογισμό των αλλιευτικών ικανοτήτων. Υπάρχουν και κοινωνικά και προβολητικά κριτήρια που θα πρέπει να συνυπολογίζονται από τους πόδα κατά την κατανομή. Δεν μα αρέσει αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη μείωση τη αλληλευτική ικανότητα, διότι προτείνει μια παγκόσμια διάσκεψη για διαχείριση που βασίζεται σε αλλιευτικά δικαιώματα για την εισαγωγή ITQs τώρα στους ε, ΠΟΔΑ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η ατραπόσε διότι αποκλείονται οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες από τα ήχθη αποθέματα ε, και θα διαπιστώσουμε συγκέντρωση σε παγκόσμιο επίπεδο των αλλιευτικών δικαιωμάτων οπότε για τις μελλοντικέ γενιές θα αποκλειστούν αυτόματα ε, κάποιες ε, χώρες και ε, θα αποκλειστεί και η αλία μικρής κλίμακας επίσης. Άλλες τώρα πτυχές για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με τα εμπορικά ζητήματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, ε, ε, ε, ιδιωτικές συμφωνίες ανάμεσα στις τρίτες χώρες και πλειοκτήτες, ε, ούτως ώστε να επικρατήσει διαφάνεια ε, στη δράση τους, να αναφέρουν τα αλλιεύματά τους στο εκάστοτε κράτος μέλος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είναι δημοσίως προσβάσιμα αυτά τα δεδομένα. Και πιστεύουμε ότι τώρα δεν μπορώ να παριθμίσω και να σας παρουσιάσω όλα τα σημεία για τα εμπορικά ζητήματα. Ξέρετε, είναι λεπτό ζήτημα, αλλά όλε οι διμερεί και πολυμερεί εμπορικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, ε, ε, υπακούν σε προηγούμενη αξιολόγηση, να ευαγούμε στου κανόνε για την περιοχή. Επίση, να εξασφαλίσουμε την ίχνη λασιμότητα των προϊόντων, ούτω ώστε να προέρχεται από νόμιμη και βιώσιμη αλία. Επίση, ο κανονισμό για την παράνομη λαθρέα και άνερχη αλία πρέπει να εφαρμόζεται. Το σημαντικό είναι οι εμπορικές συναλλαγές να μην ενθαρρύνουν, να μην μας οδηγούν ε, είτε σε υπεραλίευση είτε σε σμίκρινση των ηχθιαποθεμάτων. Στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών ε, της τη γειτονία ε, με την Νορβηγία, παραδείγματο χάρη με την Ισλανδία, πρέπει να προσέξουμε διότι ε, εκεί ανταλλάσσουμε ποσοστώσεις, ε, δεν καταβάλουμε το αντίτιμο για τα αλλιεύματα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ακολουθούμε τι ίδιες αρχές όπως και ολόκληρη η κοινιαλευτική πολιτική. Αν συμφωνήσουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ε, στις μέγιστες επιτροπές αποδόσεις τα αποθέματα ακριβώς πάνω ή, ίσε με τα, με, με τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, θα πρέπει λοιπόν να ισχύουν τα ίδια κριτήρια σε όλες τις συμφωνίες. Αυτό το θέμα δεν το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και θέλω να ακούσω ε, και τη γνώμη των συναδέλφων και παρακαλώ να ε, υποβάλλετε τροπολογίες αν έχετε ε, καλύτερες ιδέες. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να τροποποιήσουμε το κομμάτι του κειμένου που αναφέρεται σε αυτές τις βόρειες συμφωνίες. Σας ευχαριστούμε για την εξαντλητική εξήγηση. Κυρία Φράγα και κύριος Μιλάνα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, θα επεκταθώ λίγο, καθώς μου δίνετε το λόγο. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, εγώ το λέω πάντοτε ως κανόνα. Τι μου το θύμισε και η κυρία Φράγκα. Λοιπόν, αν ζητάτε από την αρχή το λόγο, πολύ καλύτερα το χρόνο. Γιατί εφόσον ε, αν δώσουμε ε, στην αρχή πολύ χρόνο στον εισηγητή και σε ήταν στην αρχή το λόγο, τότε επεκτείνονται και μετά μου ζητάτε κι άλλοι. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Γκαρσιέρο. Λοιπόν, για δύο-τρία λεπτά σας δίνω το λόγο. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ την κυρία Λεβίν ε, για την πρόταση ψηφίσματος. Δεν θα μιλήσω για τα σημεία με τα οποία συμφωνώ, αλλά θα αναφέρω που είναι οι διαφωνίες και έτσι εξοικονομώ και το χρόνο. Λοιπόν, ε, καταρχήν, έχουμε πρόβλημα με την ισπανική μετάφραση. Είναι εντελώ ακατανόητο και εγώ σε ορισμένα σημεία πρέπει να δω το κείμενο στα αγγλικά γιατί πραγματικά είναι δυσνόητο το κείμενο. Ακατανόητο λείπουν ε, κάποιες προθέσεις, υπάρχουν αλλού προθέσεις, η ορολογία δεν είναι σωστή και υπάρχουν και άλλα λάθη για το κτιμώντας ε αναφέρεται στο 208 άρθρο της συνθήκης, ενώ στην ισπανική μετάφραση λέει 201, ούτε τα νούμερα δεν έχουν σωστά. Λοιπόν, εγώ θα έπρεπε λοιπόν να κάνω μία διόρθωση στο κείμενο εδώ. Αυτό είναι το πρώτο. Βέβαια δεν την ενδιαφέρει την κυρία Λόβεν ε, γιατί είναι θέμα μετάφρασης. Τώρα, θα τα πω κάπως ανάποδα. Καταρχήν θα μιλήσω για ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, ε, που είναι στο σημείο 30, στο κτήματος ε, ό,τι αφορά ε, τα ιστορικά ελέγματα στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας. Και να σας πω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιείτε για την κατανομή των ελευτικών ε, δυνατοτήτων. Δεν είναι το μόνο σήμερα. Σήμερα όταν μοιράζουμε αυτές τις ελευτικές κανότητες της πόδα να λαμβάνουμε υπόψη και τις αναδυόμενες χώρες και ε, τις παράκτιε χώρε και δεν είναι σωστό αυτό και υπάρχει και ένα ακόμη θέμα που επίση πρέπει να έχετε υπόψη. πολλέ από αυτές τις ε, αναδυόμενε χώρε που ζητούν ε, αλευτικέ δυνατότητες ε, τις θέλουν στη συνέχεια για να τις παραχωρήσουν και έχουμε την Παππούα Νέα Γουινέα και ξέρετε τι συμβαίνει στη χώρα αυτή. Ο στόλος με τα γρηγρή έχει νέα σκάφη με δική του σημαία και πάνω από 30 σκάφη που φέρουν σημαία Παπονέας Γουισινέας, αλλά δεν είναι δικά τους. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούνται κρυφά ε, στη συνέχεια τα σκάφη αυτά και έτσι λοιπόν πάντοτε είναι καλύτερα να έχουμε κατά νου αυτή την ισορροπία. Τώρα, στο σημείο, όταν σας μιλάτε για την ε, ε, σχέση με τις άλλες πολιτικές, εγώ θα ανέφερα και το εμπόριο. Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό και το εμπόριο, πέρα από ε, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και το εμπόριο εδώ, γιατί το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή σε ελευτικά ζητήματα, όπως και το περιβάλλον και η ανάπτυξη. Και στην παράγραφο 5, όταν μιλάτε για σχέδιο δράση, διαχείριση τη ελευτικής ικανότητα, Λέτε ότι η Κομισιόν εστιάζει σε αντιφατικά σημεία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτά, γιατί η μεταρρύθμιση, στη μεταρρύθμιση θέτει τώρα ε, τα ε, μεταβιβάσιμες ε, ποσοστώσεις και το υπόλοιπο στόλος θα συνεχίζει να εφαρμόζει το σημερινό σύστημα εισόδων και εξόδων. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημείο 9, την παράγραφο 9, όταν αναφέρεστε στα Ηνωμένα Έθνη και στην ε, παράνομη λαθρεία και ανερχίαλια, δεν συμφωνώ με όσα λέτε στο σημείο 9 ε, μάλλον συμφωνώ σε αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, ε, στο ότι δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός αλίας πλά. Εγώ νομίζω ότι οι πρώτοι ένοχοι είμαστε εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια κριτική εδώ και στους εαυτούς μας και στο ότι υπάρχει έλλειψη του κανονισμού 1005 σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι και εδώ είναι αλήθεια ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι απόλυτα σαφής. Θα ήθελα να ξεκαθαριστεί ότι το, το θέμα των ε, πλεονασμάτων και παραπέμπω εδώ στη σύμβαση του ΟΗΕ και στη συμφωνία του Κατονού όπου λέγεται σαφέστατα ότι πρέπει να είναι αρμοδιότητα του τρίτου κράτους. Αυτό το κράτος που πρέπει να αξιολογήσει τα πλεονέσματα είναι αυτή η τρίτη χώρα που έχει την υποχρέωση και την αρμοδιότητα σε αυτό. Και υπάρχει και ένα θέμα που θα θέλαμε να αναφέρετε στο μέλλον, ότι τα πλεονάσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τη στιγμή τη κατανομή. Πολλέ φορέ το ευρωπαϊκό στόλο είναι ο πρώτο, ο οποίο έχει. Ε, κάποια διακριμένα δικαιώματα, επειδή είναι ο πρώτο που πήγε εκεί. Και δεύτερον, συμφωνώ με τα κριτήρια βιωσιμότητα. Ε, Πολλέ φορέ είναι ο πιο βιώσιμο. Έτσι λοιπόν, στην κατανομή των πλεονασμάτων θα θέλαμε να αναφέρονται αυτά τα θέματα. Δηλαδή, εμεί επειδή είμαστε οι πρώτοι, δεν θα μείνουμε τελευταίοι και επειδή είμαστε και οι πλέον εφόροι, δεν θα μείνουμε εκτό με μια κατανομή. Μήπω να ολοκληρώσετε, κυρία Φράγκα, πολλά μου μένουν ακόμα. Κοιτάξτε, έχουν ζητήσει το λόγο έξι άτομα. Άμα μιλήσουν πέντε λεπτά, όλοι 30 λεπτά. Λοιπόν, για την προσωρινή αλλαγή της σημαία, σημείο 14. Δεν συμφωνώ μαζί σας και θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα σαφέστατα. Στην περίπτωση της μόνο έχουμε τώρα της, ε, έχουμε μια συμφωνία που συνεχίζει να ε, εφαρμόζεται η συμφωνία αποκλειστικότητα παρά το ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο και είπατε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ε, που αλλιεύουν στην Καμπόν και ε, κλείνουν το 20% της παραγωγής της και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ικανή να δώσει διέξοδο στο θέμα αυτό, είναι κατανοητό ότι κάποιες στιγμές κάποια στιγμή θα αλλάξουν σημαία αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω. Να σας ε, πω άλλο παράδειγμα. Έχουμε ιταλικό σκάφος που άλλαξε σημαία επειδή η Ιταλία δεν επιτρέπει να έχουν ιδιωτική ασφάλιση κατά της πειρατείας και άλλαξε σημαία γιατί ήθελε να είναι ασφαλισμένο για το θέμα της πειρατείας. Δηλαδή να λέμε όχι γενικά στην προσωρινή αλλαγή ίσως είναι υπερβολικό. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα τα πω σε εσά γιατί μου μένουν πάρα πολλά ακόμη να πω και δεν πρόλαβα. Κοιτάξτε, εγώ δεν ε, είμαι σκιώδη και δεν έχω πολύ μεγάλη δυνατότητα να μιλήσω με την κυρία Λέβεν, αλλά τέλο πάντων, ο κύριο Μιλάνα. Λοιπόν, τα πράγματα για τα οποία εγώ ε, δεν συμφωνώ, θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ καλή δουλειά σας. Ε, παρόλα αυτά θέλω όμως ε, να προτείνω μια αξιολόγηση κάτι, για κάτι που λείπει και λείπει και στην πρόταση της Κομισιόν και στην ίδια την έκθεση. Και είναι το εξής, αυτή η ιδέα ότι η εξωτερική διάσταση ε, να περιορίζεται στο να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των εφιστάμενων αναλυτικών συμφωνιών. Εγώ θέλω να προτείνω μια ε, διαφορετική σκοπιά στην συγκήτρια, κάτι πολύ απλό. Στην Μεσόγειο εμείς έχουμε ένα πρόβλημα ότι η δική μας εξωτερική διάσταση είναι ε, η μοναδική πολυπλοκότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα που αφορά όλη τη Βόρεια Αφρική και αφορά και τις σχέσεις με την Τουρκία και με τη Ρωσία στον Αξινοπόντο και δεν ε, υπάρχει αξιολόγηση ε, πέρα από μια γενική έκκληση που μπορεί να απευθύνεται στο να ασχοληθούν με αυτό το θέμα οι διεθνείς συμφωνίες. Και τώρα, ε, καθώς ε, με παραδοσιακό τρόπο ερμηνεύουμε μια αλληλευτική συμφωνία, ότι είναι μια εμπορική οικονομική συμφωνία, υπάρχει όμως ε, και μια άλλη συνιστόσα κοινωνική σε μια αλληλευτική συμφωνία και υπάρχει και ένα στοιχείο αηφορίας, βιωσιμότητας. Η ερώτησή μου είναι εμείς ε, είμαστε, θέλουμε μια ιδέα διεθνών συμφωνιών που να θεωρείται μόνο ως μια δυνατότητα αλίας ε, του δικού μας ε, στόλου, των δικών μας σκαφών. Ή η μεταρρύθμιση μπορεί να εισαγάγει μια αξιολόγηση στην οποία η ελευτική συμφωνία θα ε, σχεδιάζεται και ως λύση σε μία σύραξη και στην εφαρμογή της ίδιας της πολιτικής, της αηφορίας και της διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό λείπει. Λείπει και στο έγγραφο, αλλά λείπει και στην έκθεση. Και θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το εισαγάγουμε. Ουσιαστικά προβλέπουμε εδώ ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσαν ε, να δημιουργηθούν, ε, να συναυτούν συμφωνίες ε, αλίας με τρίτες χώρες, όχι απαραίτητα εκεί όπου η οικονομική πτυχή της συμφωνίας είναι η πιο σημαντική, αλλά η αξία της εφορίας και της συνδιαχείρισης του θαλάσσιου χώρου να λαμβάνει μεγαλύτερη θέση, να είναι πιο σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, είναι διεξοδικότατη η έκθεσή της. Επιτρέψτε μου να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, ε, στην παράγραφο 10 έχω δυσκολίες, αμφιβολίες ως προς την κατανόηση. Έχω την εντύπωση ότι μετατίθεται η κοινή αλλιευτική πολιτική Μιλάμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση ή για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των ωκεανών. Φαίνεται ότι μας απασχολεί μια ενοποιημένη, μια παγκόσμια πολιτική όπου θα χρησιμοποιηθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό εννοείται. Θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε. Κατόπιν, στην παράγραφο 14... Όταν ε, απαγορεύει ετεροχρονισμένη μετανιολόγηση για να επιστρέψει ένα πλοίο στο στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε κάποια ε, στιγμή είχαμε συζητήσει να προβλεφθεί και συγκεκριμένη περίοδος, όχι απλώς μια τελεσίδικη, απόλυτη απαγόρευση. Στην παράγραφο 17 τώρα. Συμφωνώ βεβαίως, αλλά αναρωτιέμαι αυτή η δήλωση που κάνουμε εδώ δεν πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στη συμφωνία. Δεν πρέπει να αναφέρεται ρητά στη συμφωνία. Ε, και να μην εμφανίζεται με κάποια άλλη μορφή στην προκειμένη περίπτωση σαν εκτιμώντας. Ε. Κατόπιν, ε, παράγραφος 21. Μιλάμε εδώ για εξωτερικούς ανεξάρτητους ειδικού ε, που θα κληθούν να ε, κάνουν τις αξιολογίες. Επί της αρχής μπορώ να συμφωνήσω, θα ήθελα όμως να μου εξηγήσετε ποιος θα πληρώσει την αμοιβή αυτών των ε, εξωτερικών ειδικών. Από ποιο κονδύλι του προϋπολογισμού δηλαδή θα αποζημιωθούν. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η τεχνογνωσία. Τέλος, παράγραφος 26. Και πάλι μπορώ να συμφωνήσω επί της αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ηγηθεί της ενδυνάμωσης των πόδων κτλ. Όμως πιστεύω πως με κάποιο τρόπο θα πρέπει ξέρω, να προσθέσουμε ένα αντεπιχείρημα. Δηλαδή, ναι μένει να αναλυφθεί αυτός ο ηγετικός ρόλος, αλλά οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωση ε, να μην οδηγούν σε μειονέκτημα και άδικη μεταχείριση των οικονομικών φορέων τη Ένωση σε σχέση με τους εξωτερικούς φορείς, γιατί αλλιώς ε, από μόνοι μας θα δημιουργήσουμε προβλήματα στην ευρωπαϊκή αλία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αντισταθμίσουμε αυτό το επιχείρημα με μια ε, με ένα αντεπιχείρημα, όπως σας το περιέγραψα τώρα. Σας ευχαριστούμε, η κυρία Γκαρθία Ιερό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν σας άκουσα ότι είχατε πει ότι έπρεπε να ζητήσουμε το λόγο πριν να τοποθετηθεί η συγγήτρια. Σας ζητώ συγγνώμη, είναι και θα πολύ σύντομα, γιατί πράγματι αυτό σας επιτρέπει να διαχειριστείτε καλά και το χρόνο. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε τον ίδιο χρόνο, να μας δίνει σε όλους ε, τον ίδιο χρόνο. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ καλή έκθεση αυτή και θέλω να συγχαρώ την συγκήτρα και για τους στόχους που θέτει, αλλά και για την φιλοσοφία που ακολουθεί. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και είναι το κείμενο αυτό σε ό,τι αφορά μια σειρά μέτρων που εφαρμόζουμε και εμείς τους εαυτούς μας και θεωρούμε ως το ελάχιστο και που συζητούμε και θέλουμε να τα συμφωνήσουμε και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινής ελευτική πολιτικής, αλλά πρέπει να θέτουμε και σε τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν, προς αυτήν την κατεύθυνση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρονται και να κάνουμε μία πρόταση προς το να ενσωματεθούν και στα πλαίσια σύννεψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, έτσι ώστε στο μέτρο δυνατούν όχι μόνο να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, αλλά να προωθήσουμε και την ευημερία όλων των πολιτών. Κυρίως ε, γιατί η αλία σε αυτές τις τρίτες χώρες γίνεται εκεί όπου οι ντόπιοι έχουν ε, τις μεγαλύτερες δυσκολίες ε, να ζήσουν από αυτούς τους σπόρους και υποστηρίζω την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά γιατί αυτά τα δύο συνδέονται στενά. Το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Ε, το θαλάσσιο περιβάλλον ε, πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν ε, όλο ένα και περισσότερες δυσκολίες γιατί εμείς που είμαστε και κύριοι καταναλωτές και όλο και περισσότερο ε, απαιτητικοί να δεχόμαστε όταν παραδείγματο χάρη συζητάμε για την ετικέτα και για το ποιε πληροφορίε πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή, θα είναι όλο ένα και πιο δύσκολο λοιπόν να συμφωνήσουμε. Θέλουμε ως δυνατόν να καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη διαφάνεια. Αν ε, μπορείτε, θα ήθελα να με διευκολύνετε ή εσείς ή ε, Κομισιόν για το εξή. Αναφέρεται εδώ η δυσκολία που έχει η Κομισιόν να λάβει κάποιες αληθείς πληροφορίες που να μπορούν να επαληθευτούν σχετικά με το ότι πολλά σκάφη που χρησιμοποιούν τις μέτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούν αυτές τις πρακτικές. Και μάλιστα οι πληροφορίες αυτές δεν δίνονται από τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεμελιώδες, αυτό το θέμα να συγκεκριμενοποιηθεί στην αμεταρρύθμιση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη, όποια και είναι αυτά, που δεν ε, χορηγούν αυτές τις πληροφορίες για να μπορεί να γίνει μια ορθή αξιολόγηση να λάβουν μέτρα τέτοιου είδους έτσι, ώστε να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα δηλαδή από, τον, ε, από τη μαύρη λίστα μέχρι και την επιβολή κυρώσεων. Γιατί, γιατί αυτό με οδηγεί στο να σκεφτώ το εξή ότι ε, αν υπάρχουν πολλοί που αλλιεύουν υπό σημεία Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτε χώρε και δεν σέβονται του κανόνε ε, και υπάρχει επικάλυψη με την παράνομη αλλία και με την ε, αδήλωτη αλία, με τη λαθρέα αλία, τότε αυτό έχει μεγάλε επιπτώσει γιατί λέμε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος, ε, δεύτερος μεγαλύτερος οικονομικός παράγοντας που ε, προωθεί την παρανομία και την έλλειψη συμμετοχή ε, στην ανάπτυξη και των κρατών μελών αλλά και των υπόλοιπων χωρών. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, η Μεσόγειος δεν ε, μιλάμε μόνο για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι στη Μεσόγειο. Παρ' όλα αυτά, ε, κατανολώνουμε τα προϊόντα τους χωρίς να υπάρχουν ε, ίδιες εγγύσεις για τα προϊόντα αυτά που αλλιεύονται. Αν είναι δυνατό, θα ήθελα να μου πείτε αν θα υπάρχει κάποιο άλλο πλαίσιο συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Και μπορώ να σας πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ καλή έκθεση και θαραλέα, γιατί αναφέρεται στο μέχρι που μπορεί αυτή η απάτη να φτάσει, δηλαδή μπορεί να στηριχθούν και κάποιες εγκληματικές οργανώσεις, εγώ νομίζω ότι εδώ η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και να αξιολογήσει τις ε, αλευτικές πολιτικές. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λόβιν, διότι η εργασία της συμπληρώνει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα προσέθεσε η συγγήτρια νομίζω συμπληρώνουν τη μελλοντική αυτή αναδιατύπωση. Ως αναπόσπαστο μέρος της όλης μεταρρύθμισης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, διότι ακόμα μένουν πολλά που πρέπει να ρυθμιστούν στα θέματα των εξωτερικών συμφωνιών. Και επίσης για τη σχέση με τις χώρες εκείνες που δεν έχει διμερείς συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα χώρες της, του Ευξήνου Πόντου. Εγώ ήλπιζα η συγκεκριμένη αυτή έκθεση ή το τμήμα του κανονισμού το οποίο αναφέρεται στην εξωτερική διάσταση να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Είναι παράξενο ότι οι σχέσεις αυτές έχουν μείνει κάπως απ' έξω. Κατανοείτε τώρα το ενδιαφέρον μου μετά από την ένταξη βέβαια της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω λοιπόν να προτείνονται αποτελεσματικά μέτρα, αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης και λαθρέας αλίας. Ως κοιόδης εισηγήτρια, εγώ θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες καθώς επίσης και θα προσθέσω κάποιες διατυπώσεις για κοινέ συμφωνίες χωρών μελών με τις ε, χώρες αυτές. Ο κ. Χάγκλουντ. Ευχαριστώ πρώτα την Ισαβέλα για την ε, καλή της έκθεση και εγώ ως κοιόδης εισηγητής για λογαριασμό της ομάδας μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ ικανοποιητική η έκθεση και αποτελεί, έτσι γνωρίζουν άλλωστε και οι περισσότεροι συναδελφοί μου στην ομάδα μου, μια καλή αφετηρία για τις εργασίες μας. Έχουμε διαπραγματευτεί πολύ εντατικά εδώ στην ε, Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά. Και πρώτα σχετικά με τα δεδομένα. Λίγο μετά θα συζητήσουμε τη δική μου έκθεση, ότι δεν έχουμε δηλαδή επαρκή δικά μας δεδομένα για την αλληλεία εδώ στα χωρικά ύδατα των δικών μας χωρών. Είναι ένα θέμα που και εκεί πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε αν έχουμε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να εξασφαλίσουμε συλλογή καλύτερων δεδομένων στο μέλλον, κάτι που θα μας επιτρέψει να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα θέματα. Είναι βέβαια λίγο ακαδημαϊκή η συζήτηση για το εάν ε, τα δεδομένα που έχουμε για βάση, για ορισμένες συμφωνίες, είναι ορθά ή όχι. Γιατί έτσι δεν είμαστε βέβαιοι για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, αν είναι δηλαδή βασισμένες σε ορθά δεδομένα. Υπάρχουν ορισμένα ελάσσονα σημεία, για παράδειγμα το 21 στην έκθεση, που νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε όλοι να εξοικειωθούμε με αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να έχουμε και τις εκθέσεις και τα δεδομένα τουλάχιστον στα γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. Εγώ είμαι ήδη εισηγητής για ορισμένες συμφωνίες μόνο στα γαλλικά και δεν γνωρίζω ακόμα αρκετά τα γαλλικά για να μπορέσω να εργαστώ με τη γλώσσα αυτή. Αυτό λοιπόν ε, δεν ε, με εξυπηρετεί καθόλου. Νομίζω ότι χρειάζεται με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και μάλιστα ορισμένοι από εμά δεν μιλούν καν τι τρει γλώσσε που ανέφερα πριν. Κάτι άλλο είναι η προσωρινή ε, εφαρμογή των συμφωνιών. Όλοι νομίζω είμαστε απογοητευμένοι από το γεγονό ότι η Κομισιόν έχει την τάση να προετοιμάζει τι συμφωνίε αυτέ, έτσι ώστε αυτέ να μπορούν να εφαρμοστούν προσωρινά και εκ των υστέρων καλούμεθα εμεί να εγκρίνουμε την θέση τους σε ισχύ. Αυτό πραγματικά είναι, δεν είναι, είναι τρόπος για να εργάζεται το Κοινοβούλιο. Διότι δεν μπορούμε έτσι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η συνθήκη. Ίσως λοιπόν να περιλάβουμε κάτι και για αυτό το θέμα στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, νομίζω ότι είναι πράγματι σημαντικό. Συμφωνώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι η διατύπωση της παραγραφικού 22 είναι σωστή Γενικά με ικανοποιεί το ότι ζητείτε περισσότερη διαφάνεια για τις συμφωνίες αυτές. Αυτό το βρήκα σωστό όταν διάβαζα την έκθεσή σας. Και ένα άλλο αρκετά μεγάλο θέμα είναι το δημοσιονομικό βάρος των συμφωνιών που θα αναλάβει ο ίδιος ο κλάδος. Διότι ήδη ο κλάδος της Αλίας πληρώνει ένα σημαντικό μέρος, αλλά και ο φορολογούμενος επιβαρύνεται σημαντικά. Και οι επιδοτήσεις καταλήγουν εν μέρη στις τσέπες ορισμένων στον αλλιευτικό κλάδο και τους κάνουν πλούσιους. Αυτό ισχύει τώρα για ορισμένες συμφωνίες. Και το ερώτημα είναι πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το μέρος της συμφωνίας που θα αναλάβει τις δαπάνες τις σχετικές δηλαδή ο ίδιος ο κλάδος. Για την παράγραφο 40 για τις τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι εντάσσεται εδώ στην πραγματικότητα το θέμα αυτό, αφού είναι έκθεση περί αλληλείας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ρυθμίζουμε τα του τραπεζικού τομέα μέσω των εκθέσεων της Επιτροπής Αλίας. Και τέλος, να μην λησμονούμε την πολύ καλή έκθεση το 2010 του κ. Κατέκ για την εισαγωγή προϊόντων αλίας και άλλων αλληλευτικών προϊόντων και να μην λησμονούμε τις καλές εκείνες αρχές τις οποίες είχαμε εγκρίνει σχεδόν ομόφωνα εδώ. Και ορισμένα από τα πράγματα εκείνα θα έπρεπε να τα βάλουμε τούτην εδώ την έκθεση. Και τέλος, γενικότερα, όταν μιλούμε για μια πιο βιώσιμη προσέγγιση απέναντι στους εταίρους μας στην Αφρική για παράδειγμα ορισμένοι λένε μα τότε θα έρθουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και θα πάρουν τα μερίδια αυτά ταυτόχρονα εάν κάνουμε πιο ορθολογικές τις πολιτικές μας αλληλευτικοί και άλλες θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε εκεί επιτόπου καλύτερα να διατηρήσουμε τα μερίδια μας χωρίς να χάσουμε αλληλευτικές δυνατότητες ταυτόχρονα ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων Μιλώ για όλες τις πολιτικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και αλλιευτικές. Αυτό βέβαια είναι μια σημαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να δώσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για κάποια σχετική διατύπωση στην έκθεση, στην σας. Αυτά εν γέννη και είμαι πολύ ευχαριστημένος όπως είπαμε, την έκθεσή σας. Ο κ. Δεπίτερ, εξ της Κομισιόν. Yes, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. επικροτούμε την ε, εισηγήτρια για την ποιότητα της έκθεσής σας. Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Αν εξετάσουμε το σύνολο των προτάσεων που έχουμε στη διάθεσή μας, διαπιστώνουμε το 70% ε, των προϊόντων στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγόμενα, προέρχονται, προέρχονται από τα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η όλη εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος ε, κυρίως εν της μεταρρύθμισης ε, της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Χαιρόμαστε που μας υποστηρίζετε και χαιρόμαστε επίσης ε, διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υποστήριξη για τα διάφορα επιμέρους μέτρα και τα διάφορα επίπεδα στα οποία επιθυμούμε να παρέμβουμε και συμφωνείτε επίσης σχετικά με το, την διάδοση των ε, πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια των περιφερειακών οργανισμών, ε, στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών, με οικονομικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Ακούσαμε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά υποθέτω ότι μπορούμε κατηδίαν και σε μελλοντικέ συναντήσεις να τα συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια για την κυρία Λόβιν. Είναι πολύ καλή βάση για την συνέχιση των εργασιών μας και τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση σας ακούσουμε την κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας. Σημείωσα όλα τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις, γιατί είναι φράγα πρώτα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω όλα τα σχόλιά σας και αν θέλετε ίσως μπορούμε να διπνήσουμε μαζί στην Γκουάμ όταν θα πάμε εκεί την επόμενη εβδομάδα ως αντιπροσωπιά. Βεβαίως αφήνω τα χαριτολογήματα τώρα, ασφαλώς θέλω να ακούσω τα σχόλια της κυρίας Φράγα. Για την ερώτηση λοιπόν της κυρίας Φράγα λέμε ότι η Κομισιόν έχει άρει τους περιορισμούς διαχείρισης της χωρητικότητας στον κανονισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι με την πρόταση για τα TFC οι, χώρε, χώρες ή τα τμήματα που εισάγουν TFC δεν θα έχουν ποσοτικούς περιορισμούς. Μόνο για τους άλλους τόλους θα ισχύει αυτό. Για την ρήτρα αποκλειστικότητας καθώς και για την αλλαγή σημαίας. Ίσως υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν ας πούμε νόμιμοι λόγοι για να αλλάξουν σημαία κάποια σκάφη, αλλά θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου ο κλάδος δεν θα έχει νόμιμους λόγους να το πράξει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μεγάλο και πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί. Για τον κύριο Μιλάνα, ο οποίος είναι απόν βέβαια τώρα, Η κοινή διαχείριση της θάλασσας, είτε στη Μεσόγειο είτε στον Εύξηνο, βέβαια, αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στο, στην έκθεση. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία των διαχειριστικών οργανισμών και στη Μεσόγειο και, στην, και στον Εύξηνο οπότε στη Μαύρη Θάλασσα. Και για τη Μαύρη Θάλασσα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος περιφερειακός οργανισμός που να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Γιατί τώρα με την Επιτροπή της Μεσογείου δεν νομίζω ότι αποδίδει η προσπάθεια. Γενική Απατράω έθεσε ορισμένες ερωτήσεις. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Για την ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των ωκεανών. Δεν ξέρω αν ίσως οφείλεται σε μετάφραση, διότι είπε η κυρία Φράγκα ότι η ισπανική γραπτή μετάφραση δεν ήταν καλή. Δεν μιλούμε για την ευρωπαϊκή, για την ε, ε, ολοκληρωμένη ε, συγγνώμη, ε, θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει ωστόσο αυτό να έρθει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και τομείς πέραν από τις εθνικές αρμοδιότητες και όλα τα μέτρα εκμετάλλευσης που γίνονται στα πελάγια, όχι μόνο για τα ψάρια, αλλά και για υδρογονάνθρακες και για ορυκτά κλπ. Ρωτήσατε επίσης κυρία Πατράου, η Ένωση να μην ανταγωνίζεται τους ντόπιου ψαράδες για τα ίδια αποθέματα. Πρόκειται ε, ε, τυπικά τουλάχιστον για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Είναι σημαντικό ωστόσο να κατασταθούν από τώρα ήδη οι βασικές αρχές και νομίζω ότι αυτές οι βασικές αρχές πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες. Τέλος, ποιος θα πληρώνει τις ανεξάρτητες αξιολογήσεις των περιφερειακών οργανισμών. Η Κομισιόν προτείνει οι ανεπτυγμένες χώρες να πληρώνουν την ε, πρόσβαση στα αλληλευτικά αποθέματα. Να υπάρχει δηλαδή μια πρόσβαση, ένα, τίμημα για την πρόσβαση. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι καλή. Υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις, το γνωρίζω αυτό. Μπορούν να αποκλειστούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μιλούμε για διεθνείς πόρους και αυτοί που πραγματικά αποφελούνται οικονομικά από την χρήση των πόρων αυτών θα πρέπει να καταβάλουν και ένα τμήμα του τιμήματος. Η κυρία Ρότοβα, η οποία έφυγε τώρα βέβαια, έκανε την πρόταση σχετικά με την Μαύρη Θάλασσα. Θα α, ήθελα πολύ να δω και τις άλλες τροπολογίες που θα υποβάλει. Α, και κυρία Φράγκα πάλι, είπατε πολύ σωστά ότι δεν επιτύχαμε ως τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουμε όλους τους στόχους του κανονισμού. Αλλά δεν έχουμε βάλει μέσα στη λίστα στους καταλόγους της παράνομης και λαθρέας αλίας όλα τα σκάφη για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες. Επομένως το θέμα της παράνομης λαθρέας και ανεξέλεγκτης αλίας είναι πολύ σημαντικό. Και ούτως ή άλλως ψηφίσαμε πέρσι έκθεση για την αλία αυτή. Και γι' αυτό δεν περιλαμβάνω τόσα πολλά στοιχεία για αυτήν την αλία στην δική μου έκθεση. Για τον κύριο Χάκλουντ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε κυρία Λεβέν. Ε, πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής σας διάταξης. Σας συγγνώμη. 26 Μαρτίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την κάθεση τροπολογιών. Είναι πολύ σύντομος ο χρόνος. Κύριε Φράγα, παρακαλώ. Εγώ λέω ότι πρέπει να βιαστούμε γιατί εγώ θα προτιμούσα να συζητήσουμε περισσότερο τα θέματα αυτά, γιατί και για το Ταμείο δεν συζητήσαμε τόσο την πρόταση ψηφισματο. Εγώ θα πρότεινα, αν συμφωνεί και η κυρία Σιγήτρια, να παρατείνουμε την προθεσμία για τι τροπολογίε να ρωτήσουμε την κυρία Σιγήτρια, και εγώ συμφωνώ ακριβώ. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο που μας περισσεύει. Ήταν μια έκθεση η οποία κινήθηκε γρήγορα και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη προθεσμία αν και η συγγήτρια συμφωνεί. Κυρία Λαβέν. Εξαρτάται από το τι σημαίνει αυτό για να δούμε και τις ε, μελλοντικέ συνεδριάσεις της Επιτροπής, αν θα καθυστερήσει συνολικά η έκθεση. Θα πρέπει να αλλάξουμε όλο το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, προσωρινό χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. 26-30 Μαΐου στη συνέχεια και Ολομέλεια τον Ιούλιο, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να το καθυστερήσουμε χωρίς να αλλάξει ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα γιατί είχαμε προβλέψει 26 Μαρτίου τροπολογίες 30 με ψηφοφορία στην Επιτροπή και κατόπιν ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Δηλαδή θα ερχόταν το Μάιο στην Επιτροπή, έχουμε επαρκή χρόνο για να το πράξουμε, μπορούμε να καθυστερήσουμε την κατάσταση τροπολογιών μία εβδομάδα, δέκα μέρες. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Κυρία Φράγκα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δηλαδή, την είδαμε τώρα την πρόταση ψηφίσματο και η μετάφραση δεν είναι καλή. Πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το βάλουμε κάτω από το χαλί, να το ξεπετάξουμε σαν να επρόκειτο ε, μια σύσταση ή μια μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί περισσότερο το θέμα αυτό εδώ. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα ήθελα. Τώρα, εγώ σε μία εβδομάδα, σε μία έκθεση που πραγματικά η μετάφραση είναι άθλια, δεν ε, μπορώ ότι μπορώ να καταθέσω τροπολογίες και να κάνω καλή δουλειά. Πρέπει να εξετάσω τις παραγράφους μία προς μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βιαστούμε τόσο πολύ για ένα θέμα που είναι τόσο πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν... τους ενδιαφέρει όλους το ίδιο, εμάς μα ενδιαφέρει πάντως ε, Και Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, να συζητηθεί μόνο μία ώρα ένα τόσο σημαντικό θέμα μία φορά. Συγγνώμη, εγώ δεν συμφωνώ. Κοιτάξτε, δεν το ξεπετάξαμε σε μία ώρα. Είχαμε δει και το, το κείμενο εργασίας. Ε, στις... Ε, το Μαρτίου δημοσιεύτηκε. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα. Τώρα ένα, να διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, Αν διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα μπορούσε να είναι στις 8 Μαΐου. Είναι αλήθεια ότι μιλάμε όχι μόνο για την κατάθεση τροπολογιών, αλλά αν ε, θέλετε να έχουμε και νέα συζήτηση στην Επιτροπή, θα έπρεπε εκ νέου να ξαναεισάγουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτό είναι πιο πολύπλοκο. Αυτό είναι το ένα. Είναι μια εναλλακτική. Άλλη εναλλακτική είναι να αφήσουμε κατά μέρου το χρονοδιάγραμμα, να μην ε, πάμε το Μάιο και επομένω όχι με πρόβλεψη για την ε, ολομέλεια του Ιουλίου και αν υπάρχει δυνατότητα να συζητηθεί σε άλλε συνεδρίε τη Επιτροπή. Ε, Ούτω ή άλλω δεν θα έχει και ιδιαίτερη επίπτωση. Κυρία Πατράω. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση που έγινε εδώ από την κυρία Φράγκα. Είναι πολύ σημαντική για να ε, συζητηθεί τόσο γρήγορα αυτό το θέμα και έχουμε και ένα νέο άγγραφο μάλιστα ενωπιών μας. Αυτό που είπε μόλις ο πρόεδρος για το ότι μπορούμε να έχουμε προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών μέχρι τις 8 Μαΐου. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, στην Συνόδο του Απριλίου ε, μπορούμε να έχουμε μία ανασυζήτηση για αυτή τη θεματική, γιατί πράγματι θα υπήρχε χρόνος ακόμη και αν δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο θα μπορούσαμε να ξαναδιαβάσουμε το κείμενο, να ξανασκεφτούμε τα θέματα αυτά και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση. Ίσως ε, να, αν δεν είναι και τόσο μακροσκελή συζήτηση, τουλάχιστον θα είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε χειρουργικά τα προβληματικά ζητήματα. Νομίζω ότι και τα δύο θα ήταν δυνατά, αλλά ο πρόεδρος σας ξέρει καλύτερα. Υπάρχει ένα αλλά πάντοτε και το αλλά είναι ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση έχει ληφθεί ήδη η απόφαση γιατί θα κάνουμε τον Απρίλιο. Δηλαδή για τον Απρίλιο είναι αδύνατον ε, ήδη να ελοποιήσουμε και να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν προβλεφθεί. Εγώ θα έλεγα αύριο οι συντονιστέ να αποφασίσουν να προτείνουν ποια θέματα έχουμε, όμως σας ε, ξέρετε ότι είναι αδύνατο να μπουν στην ημερήσια διάταξη τη συνεδρία τη Επιτροπή τον Απρίλιο. Αν το προσθέσουμε, εγώ συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να ξέρουμε ότι πρέπει να λάβουμε την απόφαση να βγάλουμε την ημερησία διάταξη άλλα θέματα. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αλλά εντάξει, α το έχουμε ξεκάθαρο. Εγώ ευχαρίστω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α θέσουμε πιθανή, ως πιθανή ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών στις 8 Μα... Μαΐου και ας ξανακάνουμε τον Απρίλιο τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν αλλάζουν οι προθεσμίες και έχουμε και χρόνο και για να το συζητήσουμε και για την κατάθεση τροπολογιών. Αν η Επιτροπή συμφωνεί, Λοιπόν, θα δώσουμε μια εντολή στου αυριανού συντονιστέ ε, ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή του Απρίλιο γνωρίζοντα ότι θα βγουν άλλα θέματα από την ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε, κυρία Λέβεν. Ε, ε, Ουσιαστικά συμφωνώ για την αναβολή της καταληκτικής ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών τώρα για την ε, ψηφοφορία, αν θα γίνει πριν ή μετά την ε, καλοκαιρινή διακοπή. Αυτό είναι που με απασχολεί. Για το θέμα της συνεδρίασης των συντονιστών αύριο, θελήσατε να καταργήσετε τη συζήτηση για τις τροπολογίες ε, για την έκθεσή μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Συνεχίζει η κυρία Λέβιν. Ναι, θα πρέπει ε, να με ενημερώσει η γραμματεία σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων στην Επιτροπή και τι ψηφοφορίε. Δηλαδή, μετά το καλοκαίρι θα ψηφίσουμε αν ε, αποφασίσουμε υπέρ τη ε, αναβολή ή όχι. Λοιπόν, για να δούμε κάτι που μάλλον δεν ήταν ξεκάθαρο. Αν διατηρήσουμε ως τελική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών την 8η Μαΐου, δεν θα άλλαζε το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα. Δεν αλλάζουν οι υπόλοιπε προθεσμίε. Δηλαδή, η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα μπορούσε να γίνει στι 30 Μαου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούλιο του 2012. Δεν θα άλλαζε λοιπόν τίποτα παραπάνω. Και μάλλον δεν με καταλάβατε καλά για τους συντονιστές. Εγώ είπα ότι αν συμφωνήσουμε ότι πράγματι για τις τροπολογίες θέτουμε ημερομηνία στις 8 Μαΐου και θα κάνουμε συζήτηση στην Επιτροπή του Απριλίου, κάποιο άλλο θέμα θα πρέπει να βγει από την μερική διάταξη τον Απρίλιο, γιατί δεν χωράνε όλα. Αλλά με την προθεσμία 8 8η Μαΐου δεν υπάρχει τροποποίηση στις υπόλοιπες προθεσμίες. Έγκριση το Μαΐο και όλο μέλη Ιούλιο. Εντάξει, συμφωνούμε. Παρακαλώ. Ναι. Εντάξει, συμφωνώ. Μάλιστα, αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Θα έχουμε κατάσταση τροπολογιών 8 Μαΐου και θα συμπεριλάβουμε και νέο τη συζήτηση το θέμα αυτό στην Επιτροπή του Απριλίου. Και θα δούμε ποια θέματα θα αφαιρέσουμε από την ημερήσια διάταξη τη συνεδρίασή μα τον Απρίλιο. Σημείο 6 και να κινηθούμε γρήγορα γιατί έχουμε καθυστερήσει και στι 5.30 θα έρθει και επίτροπο ορισμένα μέτρα κατά των χωρών, επίση επιτρέπουν την εξαγωγή μη βιώσιμη αλεία με στόχο τη διατήρηση των αποθεμάτων. Όπω ε, ξέρετε, το Φεβρουάριο ο κύριο Γκάλεκερ μα παρουσίασε την εκθεσή του. Είχαν κατατεθεί και 14 τροπολογίε. Θα περάσουμε λοιπόν στην παρουσίαση τροπολογιών. Έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ. Πρώτα Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις που συναντήθηκαν μαζί μου για να κατανοήσουμε όλοι καλύτερα τον επίγοντα χαρακτήρα της ανάγκης να προωθήσουμε την έκθεση αυτή ε, την οποία έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό, τις προτάσεις δηλαδή Το, το μικρόφωνο του Πρόεδρου είναι ανοιχτό και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον ομιλητή. Για να επιβάλλονται κυρώσεις σε χώρες οι οποίες είναι υπεύθυνε οι οποίες είναι υπεύθυνε για μέτρα μη βιώσιμης αλίας. Έτσι λοιπόν είχαμε έναν αριθμό τροπολογιών που ε, λάβαμε υπόψη και εγώ έχω τροποποιήσει ήδη τις δικές μου τροπολογίες για να λάβω υπόψη τις τροπολογίες των άλλων ευρωβουλευτών και έχω άλλες 13 τροπολογίες από τους αριθμούς 13-26 μπορώ να σας τα πω πολύ γρήγορα η πρώτη είναι της Ιζαβέλα και έχει σχέση με την συμπερίληψη των πόδα ε, δεν έχω καμία αντίρρηση η επόμενη είναι του Πάξης που τώρα θέλει να περιληφθεί η λέξη αναλογικός πάλι του Πάξας έχω αλλά δεν είναι, δεν είναι δυστυχώς παρόν δεν βλέπω ωστόσο να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει το κείμενο αυτό με περιορισμένο δηλαδή εμπόριο σε προϊόντα αλληλείας και αλληλευτικά προϊόντα. Νομίζω ότι το κείμενο της Κομισιόν καλύπτει εδώ το θέμα. 17. Αραν κατεκ που λέει ότι θα γίνεται ανακοίνωση, στο, κοινοποίηση μάλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το δέχομαι, γνωρίζω ποια είναι η πρόθεσή του. Μπορώ ωστόσο να αντιμετωπίσω το θέμα με νέα τροπολογία την οποία θα προτείνω για την έκθεση αξιολόγησης που αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται σε κοινοβούλιο και συμβούλιο σύμφωνα και με τη διαδικασία που ισχύει και στην τροπολογία 10 του κανονισμού 108 του 2012. Αυτά θα τα εξηγήσω και διμερώ τον κύριο Κατέκ, ότι η τροπολογία αυτή δηλαδή μπορεί να καλύψει την βασική αρχή της πρότασής του. Επίσης δεν κατανοώ πολύ καλά τα διορθωτικά μέτρα διαχείρισης, διότι νομίζω ότι η σωστή διατύπωση θα πρέπει να είναι η συμβολή στην διατήρηση αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Πάλι Κατέκ στην τροπολογία του δηλαδή όπου λέει αποδημητικά ήδη από τον Αύγουστο 1995 δεν συμπίπτουν με τα ιστορικά αλλιεύματα. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να παραμείνει πιο γενικόλογη η διατύπωση όπως είναι. Η επόμενη είναι του Όλη Κρίστενσεν και της Ισαμπέλα να δουν τι ζητεί η τροπολογία τους. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει γενική διατύπωση και να αφήσουμε το κείμενο της Κομισιόν. Και μένει η τελευταία, όπου έχω ορισμένε επιφυλάξεις, είμαι βέβαιος ότι και άλλοι θα έχουν επιφυλάξεις. Η χώρα που παραβιάζει λοιπόν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαντά μέσα σε τέσσερις μήνες αυτή στιγμής λάβει την κοινοποίηση. Όχι, όχι, είναι υπερβολικά μακρό το περίοδο, η περίοδος. Εάν πάει ε, στο επόμενο, θέλει το εξαμήνου στο Συμβούλιο και είναι άλλοι τέσσερις μήνες μετά, χάσαμε όλο το περιθώριο που θα μας έδινε κάποια όθηση, ενώ θέλουμε να είναι πολύ ταχύτερα τα πράγματα για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη αλία όπως είχαμε και στο παρελθόν. Εγώ θα προτείνω λοιπόν να μπορούν να απαντήσουν στην κοινοποίηση μέσα σε ένα μήνα αυτή τη στιγμή θα την λάβουν. Γιατί τέσσερις μήνες είναι υπερβολικά μακρά περίοδος. Αυτές είναι λοιπόν οι παρατηρήσεις μου σχετικά με τις τροπολογίες. Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Και νομίζω ότι στη Σύνοδο του Συμβουλίου υπήρξε μεγάλη υποστήριξη εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ η εφαρμογή των κυρώσεων αυτών. Αλλά το πολιτικό μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και αυτά που θα πούμε εμείς και η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Και ελπίζω ότι θα έχουν κάποια ας πούμε επιρροή με τον τρόπο αυτό στις χώρες που παραβιάζουν. Τρία άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο οπότε θα μιλήσω εξ ονόματός του. Και θα ήθελα να μιλήσω σου ειδικά, αλλά τα έχει γράψει στα αγγλικά αλλά θα, θα διαβάσω τι μου έγραψε. Οι σοσιαλιστές ε, υιοθετούν και αυτή την ε, ε, πολιτική για να έχουμε βιώσιμη αλία ανά τον κόσμο. Γι' αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσει τα απαιτούμενα μέσα στις σχέσεις με τρίτες χώρες, κυρίως όταν αλλιεύουν με τέτοιο τρόπο αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να οδηγούν σε υπερβολική αλίευση και αν δεν συνεργάζονται να λαμβάνονται μέτρα κοινή διαχείρισης. Παρόλα αυτά, ε, οι σοσιαλιστές θεωρούν ότι τα μέτρα που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα με την ε, συμφωνία ίδρυσης ε, του ΠΟΕ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Θα ήταν ιδιαίτερα ατυχές να εγκρίνουμε πρώτα μέτρα και συνέχεια να ανακαλύψουμε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν διότι δεν συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο. Επιπροσθέτως πιστεύουμε ότι αν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κρατών που δεν αλλιεύουν με ε, βιώσιμο τρόπο θα πρέπει να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέτοια μέτρα αν ε, δεν ε, συμμορφώνεται με αυτά τα κριτήρια βιώσιμας αλλία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο και πρέπει στο μέτρο του δυνατού να υπάρχει αμοιβαιότητα σε αυτά τα μέτρα. Υποστηρίζουμε την τροπολογία 13 των πρασίνων προς αυτή την κατεύθυνση για να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα μέτρα μέτρα δεν χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να συνιστούν διακριτική μεταχείριση κατά κάποιων χωρών. Χρειάζεται μια πρώτερη αξιολόγηση των μέτρων από περιβαλλοντική, κοινωνική και εμπορική πλευρά και των επιπτώσεων που υπάρχουν επί των τρίτων χωρών. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε τροπολογία 16 των φιλελευθέρων και 17 του ΕΛΚ και το εκτιμώντα 8 καθώς και την τροπολογία 25 των φιλελευθέρων για το άρθρο 5. Επίσης μπορούμε να εξετάσουμε την τροπολογία 2 στη γνωμοδότηση δηλαδή, της Επιτροπής Ανάπτυξης όπου ζητούνται αυστηρότερα κριτήρια ως προς την πρώτερη αξιολόγηση αφετέρου Όμω έχουμε ε, προβλήματα σε σχέση με τροπολογία 26 που συνδέεται με το άρθρο 6. Γιατί χρειαζόμαστε καταληκτική ημερομηνία για να απαντήσει μια τρίτη χώρα στην κοινοποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Γιατί πρέπει να είναι ακριβώ τέσσερι μήνε η περίοδο αυτή. Ε, οι τροπολογίε 15 και 18 του EFD δεν είμαστε σίγουροι ε, αν όντω συμβάλλουν στο να γίνει πιο ευανάγνωστο το κείμενο, ούτε και διευκρινίζουν ποιε είναι οι επιπτώσει αυτέ οι τροπολογίε και κατά τη γνώμη μα θα έπρεπε να εξεταστούν περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκαλακέρ για την εκθεσή του. Θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε ο κύριος Παντεκόπ ε, στο τελευταίο τμήμα ε, των εισαγωγικών του παρατηρήσεων για το χρόνο γιατί εδώ ο χρόνος, το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, όλοι ε, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα χωρίς να λέμε σε τι αρχικά ε, σκόπευε, δηλαδή ε, στο ότι η Ισλανδία και οι Φαρόες, και οι Φαρόες ήθελαν να αρχίσουν, ε, θέλουν να αρχίσουν τον Ιούλιο φέτος αυτή τη μακροαλίευση, θα είναι ο, το τρίτο έτος ε, που στοχεύουν ε, στο στο Σκουμπρί έχουν θεσπίσει 150.000 ε, τόνους στο στόχο και δηλαδή ε, αυτό σημαίνει ότι θα σκοτώσουν ένα εκατομμύριο τόνους του Σκουμπριού ενώ είχε πει το Επιστημονικό Συμβούλιο ότι με αυτόν τον τρόπο τίθεται σε κίνδυνο ε, η βιωσιμότητα του αποθέματος ε, και δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε να συνάψουμε κάποια συμφωνία με τη Ισλανδία και τις Φερόες τώρα και έτσι θα αφαιρέσουν αυθαίρετα αυτό το απόθεμα, αυτό το τμήμα του υποθέματος ε, και είναι σημαντικό να φροντίσουμε να το προλάβουμε για το χρόνο. Και γι' αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό και σε τέσσερις μήνες είναι εντελώ αδύνατο. Ε, αν ε, πετύχουμε αυτή την προθεσμία, ένας μήνας ε, είναι σημαντικός και πρέπει να θυμόμαστε για την Ισλανδία ότι εισάγουμε από αυτούς περίπου ε, ψάρια αξία ενό δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, κυρίως προσφυγάκι και γάδο και πολύ λίγο σκουμπρί και ε, θετώ υπόθηκαν από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες να είμαστε προσεκτικοί να μην ε, παραβιάσουμε τους κανόνες του ΠΟΕ. Όμως, ε, σε σχέση με τις Φαρόες, Έχουμε πολύ μεγάλα ενδιαφέροντα των Ολλανδών, ε, δηλαδή για να χτιστεί ένα νέο εργοστάσιο για την επεξεργασία, τη μεταποίηση του σκουμπριού. Μπορούμε να, λάβουμε, να εφαρμόσουμε κυρώσεις κατά των ίδιων των κρατομελών, να τους απαγορεύσουμε να συνεργαστούν με κάποιους που αλλιεύουν έτσι παρανόμως και ε, πραγματικά αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν ε, παραβιάζει απόλυτα ε, τις συμφωνίες με τα παράκτια κράτη. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν τον ε, Πατικοπ Γκάλεκερ και πρέπει να δράσουμε στο δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ κυρία Λέβεν. Uh, very much. thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλαχερ υποστηρίζουμε τις προτάσεις και οι τροπολογίες ε, που αποσκοπούν στην διευκρίνηση του ότι όσα αποθέματα αποτελούν αντικείμενο διαχείριση από τους πόδα έχουν από αυτή την πλευρά ιδιαίτερη σημασία και άρα ε, πιστεύουμε πως ε, είναι πολύ ε, καλή αυτή η πρόταση και θέλω να ευχαριστήσω την Ισλανδία για τα όσα έκανε διότι ε, εκείνη έθεσε το ζήτημα επιτάπητος και έτσι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι είναι θέμα διατήρησης αποθέματος και όχι εμπορικό ζήτημα. Πρόκειται για ε, πόρους που ανήκουν σε όλους και πρέπει να διαχειριστούμε σε διεθνές επίπεδο και άρα είναι θέμα διατήρησης του αποθέματος και καμία σχέση δεν έχει με παραγωγή αγαθών που εμπορευόμαστε. Είναι εντελώς διαφορετική ε, κατάσταση όταν μιλάμε για προϊόντα και θα ήθελα να εφαρμοστεί αυτό. Σας ευχαριστούμε η κυρία Φράγα τώρα. θα ήθελα να σας πω... Ότι συμφωνώ με τον κύριο Γκάλαχερ και τον ευχαριστώ που περιέλαβε τα θέματα στις τροπολογίες του, αυτά δηλαδή που είχα ζητήσει εγώ. Όντως είναι, όπως είπε και ο ίδιος, ένα εξαιρετικό όπλο για εξαιρετικές περιστάσεις. Και βέβαια πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ λοιπόν εν τέλει με τον κύριο Γαλαχρή και τον ευχαριστώ για την συνεργασία του. Thank you. Thank you for the uh, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Δύο σύντομα σχόλια. Η Κομισιόν συμφωνεί σε ό,τι αφορά την ανάγκη ταχείας υιοθέτησης του μέτρου για τους λόγους που αναπτύχθηκαν άλλωστε σαφώς εδώ Πιστεύουμε επίσης ότι και το Συμβούλιο συμφωνεί. Ελπίζουμε ότι αυτή η νομοθετική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα για προφανείς λόγους. Το δεύτερο σχόλιο μου έχει νομικό χαρακτήρα. Είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να είναι αποτελεσματικά και να έχουν πράγματι το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εμπορίου και κυρίως της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, του ΓΚΑΤ. Η νομική γνωμοδότηση που λάβαμε όταν υποβάλαμε την πρόταση ήταν ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν εξαντλεί τα όρια της νομιμότητας υπό τους όρους του ΓΚΑΤ. Το λέω αυτό για να εγγραφεί στα πρακτικά και ε, αναφέρομαι εμέσως σε ορισμένες τροπολογίες. Είναι δηλαδή σκόπιμο να εξεταστεί πολύ προσεκτικά η συμβατότητά τους με τις διεθνείς διατάξεις. Ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει σχέση με την διατήρηση ενός είδους, ενός αποθέματος κοινού ενδιαφέροντος. Και πρέπει να περιοριστεί και να οριστεί το πεδίο εφαρμογή των μέτρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν σε ενδεχόμενο έλεγχο από πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτό το σχόλιο ήθελα παρακαλώ να λάβετε υπόψη. Κύριε Γκάλαχερ, για... έχετε το τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους της Επιτροπής μας για, την... για τις παρεμβάσεις τους. Βεβαίως, με ιδιαίτερη χαρά θα περιλάβω τις απόψεις των συναδέλφων, των σκιωδών, εισηγητών ιδίως. Φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά απόψεων για τους τέσσερις μήνες. Νομίζω όμως ότι ο ένας μήνας είναι λογική υποθυσμία και για αναφορά στην ΓΑΤ κοιτάξτε, θα είμαι κοινικός. Εάν είχαμε δεχτεί την πρόταση της Κομισιόν χωρίς να την τροποποιήσουμε καθόλου. Θα μπορούσα να βγω κοινικά και να πω ότι οι Ισλανδοί έχουν αντιδράσει. Μα τότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, διότι 95-98% του Ισλανδικού σαφριδιού πουλιέται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Τότε λοιπόν θα ψάξουν να βρουν μια αγορά για τα υπόλοιπα 2-3% που μένουν. Το ζήτημα είναι η Κομισιόν μπορεί να προβλέψει κάτι εντονότερο, κάτι ισχυρότερο, γιατί εδώ μιλούν για αναπολεσματικά και για την ανάγκη συμβατότητας. Αναβρεθεί τότε κάτι που να είναι πιο αποτελεσματικό. Έχω σεβασμό για την άποψη του αξιωματούχου της Επιτροπής, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι κάτι το αποτελεσματικό. Και η δική μας νομική υπηρεσία γνωμοδότησε και μας είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και ξέρω από αυτά που είχε πει ο Στρόαν Στίβενσον και άλλοι ότι οι ποιε θα είναι οι επιπλοκές από, για άλλες χώρες που εισάγουν άλλα είδη. Ελπίζω να μην χρειαστεί ωστόσο να επιβληθεί το μέτρο αυτό. Όλοι είμαστε όριμοι άνθρωποι και θα δούμε τότε. Μα οι Ισλανδοί οι Φερόες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι κάθονται από μακριά και κοιτούν. Δεν θέλω βέβαια να γίνει. Δεν θέλω να φτάσουμε να κάνουμε και πόλεμο. Εάν η Κομισιόν, η Νορβηγία δεν πρόκειται να αναλάβουν την πρωτοβουλία, ε, τότε φοβούμε πολύ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για να λύσει το πρόβλημα. Ίσως να κάνουμε το πρώτο βήμα αυτό και να συναντηθούμε τους Ισλανδούς την επόμενη μήνα, την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Όλοι έχουμε ταχθεί υπέρ μια βιώσιμη αλληλεία για το συμφέρον των μελλοντικών γενιών και δεν καταφέρνουμε να λύσουμε ένα ζήτημα βιωσιμότητα των ψαριών για τούτη την εδώ τη γενιά, για την παρούσα γενιά. Και οι μελλοντικέ γενιές οι οποίες θα εξαρτώνται από τα αποθέματα του Βόρειου Ατλαντικού ή του Βόρειο Ατλαντικού, Ατλαντικού θα δουν ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτές. Μιλούμε για την σημασία των απορρίψεων στη θάλασσα και όλες τις άλλες σχετικές εκθέσεις και εδώ κοιτάμε, δεν κοιτάμε τα του σπιτιού μας. Να κάνουμε κάτι το οποίο είναι δυνατόν να πετύχει μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Το μόνο που λέω είναι αυτή, αυτό είναι το πολιτικό μας μήνυμα, μια πολιτική δήλωση. Θεωρούμε ότι έχουμε νομική βάση για να κάνουμε τη δήλωση αυτή. Δεν θέλουμε καθυστερήσει σε κανένα επίπεδο, ούτε από την Κομισιόν ούτε από το Συμβούλιο διότι εγώ δεν πρόκειται να συμφωνήσω ξανά. Αλλά δεν ξαναμπαίνω σε ιστορίες μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης σε τέτοια περίπτωση. Τι νόημα έχουν τα μακροπρόθεσμα ε, σχέδια διαχείρισης όταν δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα του σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό που με απασχολεί είναι αυτή η βασική αρχή. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο χωρίς να χρειαστεί να καταλήξουμε στα όπλα. Λέει είναι μαχητική οι Ισλανδοί. Α, δεν έχετε δει εγώ πόσο μαχητικός είμαι. Θα πάω την επόμενη εβδομάδα. Μήπως εκεί ο πρόεδρος χρειαστεί να ζητήσει κάποια προστασία. Καλά, στη χειρότερη περίπτωση θα φέρουμε τη φράγα. Ευχαριστώ κύριε Καλαγιάννη. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ζητήσετε προστασία. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο αυτό υποχρεώσει κοινοποίηση που προέρχονται από τον κανονισμό 2371 για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελευτικών πόρων δυνάμει τη κοινή ελευτική πολιτική. Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση και το λόγο έχει ο κύριο Χάγκλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, έχουμε ήδη συζητήσει κάποιες φορές την έκθεσή μου, οπότε θα ήθελα να τη διατρέξουμε εντάχει. Ούτως ή άλλως μίλησα λίγο για αυτή όταν σας παρουσίασα τις προθέσεις μου ε, για αυτή την έκθεση. Ε, βασιζόμαστε σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για την ε, βιώσιμη εκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων βάσει της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Αυτή είναι η βάση ε, για την έκθεσή μου. Επίσης, επέλεξα ε, να ε, ρίξω το βάρος σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Μπορούμε να τονίσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι το 60% των αποθεμάτων αλλιεύονται πέρα από το MSY, ε, την μέγιστη βιώσιμη απόδοση δηλαδή. Θέλω να το τονίσουμε αυτό. Επίσης το θέμα των ποσοστώσεων έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αποτελεσματικό για την βιώσιμη ε, μακροπρόθεσμη διαχείριση των αλλιευμάτων, Το μακροπρόθεσμα αλλιευτικ... προγράμματα αλλιευτικής διαχείρισης είναι η σωστή ε, λύση. Επίσης έχουν χαθεί πολλές θέσεις απασχόλησης στον κλάδο τα τελευταία χρόνια κυρίως επειδή ε, τα ηχθιαποθέματα είναι σε κακή κατάσταση και έχουμε πάρα πολλές και φθηνέ εισαγωγές από άλλα μέρη του κόσμου. Επίσης με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις εξή. Ε, αυτόματα έπρεπε κάποιοι να εγκαταλείψουν τον κλάδο και ε, να αφήσουν αυτή τη δουλειά σε νεότερου. Επίσης, σε σχέση με την ε, έκθεση της κυρίας Λεβίν και την ανάγκη για αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μελλοντικά θα χρησιμοποιούνται, θα έχουμε τέτοια αξιόπιστα δεδομένα και θα χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη αποφάσεων ε, σχετικά με την αλληλευτική ικανότητα, σχετικά με το στόλο, σχετικά με το απόθεμα κάθε ψαριού. Δεν μπορεί να μας ζητούν να λαμβάνουμε σοβαρέ αποφάσει χωρί να έχουμε μεριμνήσει την μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, ότι εν τέλει θα έχουμε όλα τα απαιτούμενα δεδομένα. Ε, το αναφέρω σε διάφορα σημεία, κάνω κάποιες ενθαρρυντικές προτάσεις και κάποιες σκληρότερες προτάσεις. Σε κάποιες ε, περιοχές έχουμε προβλήματα με τις φώκες, τα θαλασσοπούλια, ε, και ω προ την κατάσταση των αποθεμάτων σε κάποιε περιοχέ ε, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, ενώ σε άλλε δεν είναι, το αντιλαμβάνομαι. Uh, Γενικά τονίζω ότι τα μακροπρόθεσμα ε, προγράμματα διαχείρισης που πρέπει να ακολουθήσουμε ε, ε, η οικοσυστημική προσέγγιση είναι το κεντρικό ε, στοιχείο αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα αναφέρουμε, αλλά είναι η πρώτη φορά που το διευκρινίζουμε μέσα σε έκθεση. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι αλληλεί πρέπει να δεχτούν τον έλεγχο των αλλιευμάτων. Harvest control, όπω είναι γνωστό ε, στα αγγλικά. Σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση πρέπει να εμπλακούν ε, έτσι περαιτέρω οι περιφερειακοί γνωμοδοτικοί οργανισμοί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων ε, προγραμμάτων ε, διαχείρισης. Επίση, τοποθετούμε σε σχέση με την ε, πολιτική για τις Ε, Έχουμε συζητήσει πολλά στο θέμα και ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη ω προς αυτό η Επίτροπος. Ε, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και αυτό σχετίζεται άμεσα και με την ε, κατάσταση των αποθεμάτων. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως η πολιτική απορρίψεων θα πρέπει να βασίζεται στα αλλιεύματα και όχι στα επιμέρους είδη. Ε, ας επανέλθω τώρα στο θέμα των αξιόπιστων δεδομένων το θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε όλα τα κράτη-μέλη να αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα αξιόπιστα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν ω αίρισμα για την ε, λήψη αποφάσεων. Κάποιοι έχουν ε, πολύ καλέ επιδόσει ω προ την ε, προσκόμιση στατιστικών δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ποια περαιτέρω θα αναλυφθούν για να αντιληφθούν πρώτα τα κράτη-μέλη τη σημασία των αξιόπιστων δεδομένων και στη συνέχεια να τα προσκομίζουν. Ω προ τι αλλιευτικέ ικανότητε, τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα της υπεραλίευσης. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για όλους ότι δεν έχουμε έναν ικανοποιητικό ορισμό για την ε, υπερβάλλουσα αλλιευτική ικανότητα και τι συνιστά ε, βιώσιμο επίπεδο είναι επίσης κάτι που δεν έχουμε παρκώς ορίσει και άρα θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση, ε, βιώσιμο επίπεδα ανακράτως, αυτό πρέπει να ορίσουμε και την υπερβολική αλλιευτική ικανότητα. Επίση, θα πρέπει να εξεταστεί το τι χρειάζεται να κάνει το κάθε κράτο μέλο, λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στα οποία η Αλία είναι ε, πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με την κατάσταση πριν από 15 και 20 χρόνια. Ε, ε, δεν είναι μεγαλύτερος ο στόλος, είναι πιο αποτελεσματικός, μπορεί ε, να μην είναι μεγαλύτερα τα σκάφη παραδείγματο χάρη του στόλου αλλά είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τι μεταβάσιμες ε, αλλιευτικέ παραχωρήσει. Είναι πάρα πολύ ε, λεπτό το θέμα και κάποιοι είναι κατά του συστήματο. Πάντως αυτές οι μεταβάσιμες παραχωρήσει τα TFCs είναι ένα μέτρο που θα μα βοηθούσε να καταπολεμήσουμε την υπερβολική αλλιευτική ικανότητα αλλά δεν είναι το μόνο. Όταν μια χώρα μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει υπερβολική αλλιευτική ικανότητα και μπορεί να βρει κάποιο κάποιο άλλο τρόπο να διαχειριστεί ε, το πρόβλημα αλληλευτικής ικανότητα. δεν θα έπρεπε εμεί να επιβάλλουμε αυτό το υποχρεωτικό σύστημα των TFC. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να, ε, να λαμβάνονται υπόψη οι, ε, οι εναλλακτικέ λύσει. Σίγουρα τα TFC είναι ένα καλό τρόπο καταπολέμηση υπερβολική αλληλευτική ικανότητα. Σχετικά με τα ύδατα τα 12 μίλια, η πρόσβαση που ίσχυε δηλαδή για πολύ καιρό Πιστεύω ότι είναι καλή πρακτική και πρέπει έτσι να παραμείνει. Δεν υποβάλλω καμία πρόταση σε σχέση με αυτά. Ε, ιδού δεν πρόσθεσα και πολλά σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση και ε, θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη έκθεση πρωτοβουλίας πρωτού προχωρήσουμε σε πιο σημαντικές εκθέσεις άλλων συναδέλφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με μεγάλο μέρος του κειμένου του συναδέλφου Χάγλου σε ό,τι αφορά κυρίως το σημείο 6 όταν ε, αναφέρεται στην ισορροπία μεταξύ οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και ε, κυρίως όταν ε, αναφέρεται στην αναγκαιότητα να αυξηθεί η συμμετοχή των εκπροσώπων ε, του Περιφερειακού Γνωμοδοτικών Συμβουλίων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ε, συμμετοχή και των αλλιέων. Συμφωνώ με τον συγητή όταν ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει ορισμό για την αρισταχνική αλία για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τα μέτρα για την αλία και αυτό συγκεκριμένο τομέα εγώ προσδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στην ερασιτεχνική αλία, γιατί εκεί δραστηριοποιούνται οι οικογένειες, αλλά έχουμε και επίπτωση και στην επικράτεια. Επίσης, συμφωνώ ότι οι ε, μεταβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις δεν είναι ο μόνος τρόπος να μειωθεί το πλεόνασμα και η πλεονάζουσα ικανότητα και πρέπει να προωθηθεί και η χρήση επιλεκτικών εργαλείων. Αντίθετα, με προβληματίζει με προβληματίζουν τόσο αναφέρονται στην παράγραφο 7, όπου υποστηρίζει ο εισηγητής ότι η απαγόρευση των απορρίψεων θα πρέπει να καθορίζεται ε, στη βάση της αλευτικής δραστηριότητας και όχι σε σχέση με τα διάφορα αποθέματα, αποθέματα. Εγώ είμαι πεσμένος ότι θα μπορούσαμε να διεκδικούμε σε μείωση των απορρίψεων και και τα δύο μέτρα και επομένως δεν είναι χρήσιμο να αποκλείσουμε εδώ ε, τα αποθέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Χανλούν ότι συμφωνούμε με την προσέγγιση που ακολουθεί στην εκθεσή του. στο τέλος παρέμβασής μου θα κάνω κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια. Βέβαια, να σας πω ότι κατά την άποψή μας είναι θετικό ότι η έκθεση περιλαμβάνει τα κύρια σημεία Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων, δεν είναι μόνο λέξει κλειδί αυτέ, αλλά είναι πολύ βασικέ ιδέε που, κατά την άποψή μα, θα πρέπει να καταστούν ο πυλώνα και το κριτήριο τη νέα κοινή ελευθερική πολιτική. Απαριθμό εδώ, χωρί να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά για να είναι σαφή τα πράγματα τα σχέδια, τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης ε, που θα βασίζονται σε μια οικοσυστημική προσέγγιση, συλλογή επιστημονικών δεδομένων, απαραίτητο για να ε, έχουμε βάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση, μείωση της ελευτικής ικανότητας των στόλων σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους, ο στόχος ε, των μηδενικών απορρίψεων ε, και συμφωνούμε μαζί σας ε, στο είδος της αλίας και όχι για τα εκτεποθέματα, περιφερειοποίηση, να είναι όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη περιφερειοποίηση για την και για τη συμμετοχή των ε, Περιφερειακών Γνωματοτικών Συμβουλίων έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να οικειοποιηθούν αυτή την βιώσιμη πολιτική αλίας. Επίσης, δικαιώματα που να βασίζονται στη βιωσιμότητα αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και ε, κάποιες διευκρινήσεις ε, θα δοθούν μέσω τροπολογιών αλλά γενικά σας υποστηρίζουμε πλήρως. Ωστόσο, έχουμε δύο προβλήματα διαφορετικά στο χαρακτήρα τους ε, και ίσως ε, να καλύπτουν κάποιες αποκλήσεις. Ε, πρώτον, μερικές φορές επιμένετε στην έκθεση αυτή για το ότι βλάπτουν τα θαλασσοπούλια και οι φώκες τους ολοτικούς πόρους. Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, δεν υπάρχει ταμπού, μπορούμε να ε, αμφισβητήσουμε αυτή τη δήλωση, είναι αμφισβητήσιμη, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς ε, δεν κατανοούμε τι νόημα έχει κάτι τέτοιο εδώ στην έκθεση αυτή, μια τέτοια αναφορά. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να παραμείνει στο πλαίσιο της κοινής πολιτική και όχι να επεκταθεί και κατά την άποψή μας δεν έχει νόημα να μετακινήσετε και σε άλλα θέματα. Εμείς ε, προτείνουμε να το σβήσετε αυτό όχι για να τα βάλουμε κάτω από το χαλί και να τα καλύψουμε, αλλά γιατί θέλουμε να επικεντρωθούμε στον κύριο στόχο της έκθεσης. Δεύτερη απόκληση, πιο σημαντική, κατά την απόψή μας, το θέμα των ατομικών μεταβάσιμων ποσοστώσεων. Ξέρουμε ότι αποτελεί αυτό ένα βασικό στοιχείο της πρότασης της και συμφωνούμε, συγγνώμη, διαφωνούμε κάθετα με αυτό. Ε, πρόσεξε ότι εσείς ε, έχετε μία σόφρονα θέση. Ε, λέτε ότι είναι ένα από τα πιθανά εργαλεία, όχι ότι είναι κάτι θαυματουργό, αλλά κατά την άποψή μας και έχουμε τοποθετηθεί σχετικά. Αυτό το σύστημα των μονομένων ποσοστώσεων, των ατομικών ποσοστώσεων, είναι ένα σύστημα το οποίο ζημιώνει την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλευτικών πόρων. Ευχαριστώ, κυρία Λέβεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω λίγα μόνο στοιχεία, διότι ο συνάδελφος με πρόλαβε ε, και εξέφρασε και τη δική μου θέση. Ευχαριστούμε, Κάρλα, για την έκθεσή σου και συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό να τονίσουμε πόσο ε, σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να προσκομίζουν αξιόπιστα δεδομένα. Είναι σημαντικό που προτείνουμε να εισαγάγουμε κυρώσεις και αυτό πρέπει να κάνουμε κατά των κρατών ε, που δεν προσκομίζουν αυτά τα δεδομένα παρότι είναι επεχρεωμένα βάσει της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ε, χρειαζόμαστε δεδομένα για την αλληλευτική ικανότητα, για την εφαρμογή ε, των μέτρων και των προγραμμάτων για όλα όσα έχουμε συμφωνήσει. Επίση, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα τη υπερβολικής ε, ικανότητα. ικανότητας. Δεν υπάρχει όριο ε, για αυτήν ε, μέσα στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τη μόνη πρόταση, το μόνο όριο που έχουμε είναι τα TFC, τι μεταβιβάσιμε παραχωρήσει. Άλλο όριο δεν υπάρχει σε σχέση με τον τρόπο αξιολόγηση τη αλληλευτική ικανότητα για να μειωθεί η τελευταία και να έχουμε ένα συγκεκριμένο όριο ας πω και κάτι αρνητικό, ε, κατά τη διαστολή με τον συνάδελφο εδώ πίσω, δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό που δηλώνουμε πως χρειαζόμαστε μία ισορροπία ανάμεσα ε, στην οικονομική, κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα. Η οικολογική βιωσιμότητα είναι προϋπόθεση για τις άλλες δύο βιωσιμότητες. Ε, δεν γίνεται οικονομικός και κοινωνικός πώς να είναι βιώσιμα η εργαλεία αν δεν έχουμε ε, κρατεά αποθέματα. Θα βελτιωθεί η κατάσταση αντίθετα και η οικονομική και η κοινωνική αν είναι σε καλή κατάσταση ε, τα αποθέματά μας ε, και είναι αρκετά ζωντανά. Έχουμε ένα χωριστό ε, σύστημα για την αλία ε, μικρής ε, κλίμακας. Δεν υπάρχει συμφωνία σε σχέση με τον ορισμό, αν θα την αποκαλούμε αλία κτλ. Στη συνέχεια για τα θαλασσοπούλια δεν συμφωνούμε δυστυχώς ε, καλέ. Αυτή η έκθεση που σας έδειξα τώρα παρουσιάστηκε και στο Κοινοβούλιο και μας διαβεβαίωσαν ότι ε, ε, δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα σε συγκεκριμένα θαλασσοπούλια και τα ίδια αποθεμάτων. Θα συμφωνήσω με ε, τον ε, συναδελφό ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά μέσα στην κοινή ελευτική πολιτική γιατί μιλάμε για τα δελφίνια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που επηρεάζουν την αλία Όμω, δεν ρυθμίζονται μέσα στην κοινή ελευτική πολιτική γιατί ρυθμίζονται από άλλε πολιτικέ. σε σίγουρα, ε, σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε την κατάσταση για τα θαλασσοπούλια στη δεκαετία του 90 είχαμε 300.000 περίπου στη Βαλτική σήμερα έχει πέσει ο ρυθμός τους σε κάτω από τα 40.000. Καταλαβαίνετε ε, ότι από ιστορικής πλευράς παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός τους είναι σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση. Και εκείνοι πρέπει να φάνε και εκείνα πρέπει να φάνε. Δεν έχουν τι να φάνε και ψάρια τρώνε. Τι να κάνουμε. Αυτά ε, επιτάσσει η φύση. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε τα θαλασσοπούλια. Αυτά. Ευχαριστώ. κυρία Φράγα. Ε, λοιπόν, εγώ δεν ε, θα επικεντρωθώ στους κορμοράνους, αλλά θα κάνω μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις προάλλες, το ελεγκτικό συνέδριο ε, ενημερώθηκε σχετικά με την ε, η ικανότητα και ποτέ δεν υπήρχε ορισμός και δεν έχει γίνει ανάλυση ένα κράτο ούτε τα ίδια τα κράτη-μέλη το έχουν κάνει, ούτε υπήρξε προσαρμογή των ε, πόρων με την ικανότητα και τα λοιπά της προάλλες. Η Επίτροπος Δαμανάκη όταν συμμετείχε στην εδρίαση του ΕΛΚ είπε και εμένα με εξέπληξε αλλά όσοι τη συνόδευαν με το, μου το επαλήθευσαν ότι η Επιτροπή κάνει μία μελέτη, μία ανάλυση για το θέμα αυτό. Και εγώ θα ήθελα οι εκπρόσωποι της Κομισιόν που βρίσκονται εδώ να μας εξηγήσουν. Τι γίνεται με τη μελέτη αυτή, πώς υλοποιείται, πότε θα ολοκληρωθεί να μα δώσουν κάποιε περαιτέρω εξηγήσει σε αυτό που ανακοίνωσε η κυρία Δαμανάκη τη προάλλες, ότι υλοποιεί αυτή τη μελέτη αξιολόγηση σαν κράτο μέλο Κομισιόν σε σχέση με την τη ικανότητα. Και θα ήθελα να μα εξηγήσει η Κομισιόν ε, μία και καλή το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σπυρίλο. Απλώ θέλω να απαντήσω στη συνάδελφο, δεν μπροστά γιατί αναφέρθηκε σε αυτό που είπα εγώ. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η ισορροπία μεταξύ της οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης ε, δεν ε, είναι μόνο δική μου σκέψη. Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι και σκέψη του εισηγητή. <laughs> Το αποδώσατε σε μένα δεν είναι έτσι, αλλά εγώ συμφωνώ και νομίζω ότι είναι σωστό και συνδέεται και με το γεγονός της συμμετοχής των αλλιέων στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα για να ξεκινήσουν νέες διαδικασίες και για να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο φάκελος αυτός. Ο κύριος Παρδεκούπερ από την Επιτροπή. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την, ε, τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι εξαιρετική και καλύπτει ε, όλα τα στοιχεία που καλύπτει και η δική μας έκθεση για το ίδιο θέμα. Είναι ιδιαίτερα περιεκτική και όχι μόνο αυτό. Παρατηρήσαμε ότι πρόσθεσε κάποια στοιχεία που κατά τη γνώμη του έχουν σημασία στο, στην όλη συζήτηση. Δεν θέλω τώρα να διατρέξω όλη την έκθεση και να σχολιάσω όλα τα επιμέρους σημεία. Θα επιλέξω κάποια. Πρώτον, Πιστεύω ότι κάποιοι βουλευτές και η έκθεση τονίζουν την ε, ανάγκη να έχουμε καλύτερα και πιο αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα. Φυσικά ε, γνωρίζουμε το πρόβλημα και είναι ξεκάθαρα μια αρμοδιότητα των κρατών μελών, αυτό είναι σαφές. Τα κράτη-μέλη καλούνται να ε, που μας προμηθεύουν με τα απαιτούμενα δεδομένα επί τη βάση των οποίων διεξάγουμε και τις επιστημονικές αναλύσεις και έτσι μπορούμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Τα κράτη-μέλη πρέπει λοιπόν να παράσχουν υψηλού επίπεδου δεδομένα και γι' αυτό το στόχο χρειαζόμαστε περισσότερα, περισσότερους πόρους. Τώρα προτείνουμε αύξηση των πόρων στο Ταμείο Αλίας για να ενισχύσουμε τα κράτη-μέλη σε αυτή τους την προσπάθεια. Πάντως είναι θέμα εθνικό. Από πλευράς οικονομικής και από πλευράς προσωπικού είναι θέμα εθνικό και γι' αυτό ε, έχουμε αρχίσει ένα ιδιαίτερα εντατικό διάλογο με τα κράτη-μέλη σχετικά με την ευέλτιστη πολιτική που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ώστε να βελτιώσουμε τις γνώσεις που έχουμε, το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατάρτιση των εκθέσεών μας. Επιδιώκουμε δε ενισχυμένη συνεργασία για να βρούμε ένα πιο στρατηγικό σύστημα συλλογή στατιστικών δεδομένων και να αναβαθμίσουμε την επιστημονική βάση των αποφάσεών μας. Ε, χαιρόμαστε που υποστηρίζετε τις προτάσεις μας. Πρέπει να αναλάβουμε δράση επίσης ε, ούτως ώστε οι επιστήμονες και η βιομηχανία να συνεργάζονται πολύ περισσότερο ε, γιατί ε, καλές είναι οι επιστημονικές συμβουλές αλλά ο Αλίας είναι αυτός που καλύτερα να εφαρμόσει όλες τις επιστημονικές συστάσεις. Μόλις πάρουμε λοιπόν τα απαιτούμενα δεδομένα χρειάζεται καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην επιστήμη και τον κλάδο για να γίνει σωστή χρήση αυτών των αυξημένων και για μας είναι εξίσου σημαντικό αυτό. Θα ήθελα για την πλεονάσια ικανότητα να προσθέσω κάποια πράγματα και σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Εφράγα. Όντως, ε, πάντοτε εξετάζουμε, πάντοτε ε, εξετάζαμε αυτό το θέμα στα πλαίσια της αναθεώρησης του γενικότερου κανονισμού και αυτό συμπεριλαμβάνεται ε, εν μέρη και στην έκθεση αξιολόγησης σε όλες μας τις διαπραγματεύσεις ασχολούμαστε με το θέμα της πλεονάσας ικανότητας και επίσης επιδιώκουμε να έχουμε έναν επακριβέστερο ορισμό. Πριν από δύο χρόνια ε, η ΣΤΕΦΚΑ, αυτή η Επιστημονική, Κοινωνική και Τεχνική Επιτροπή για τα Αλλιεύματα, συμβούλευε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της ε, ε, πλεονάσας ικανότητας εμείς διαρκώς ε, ε, ζητούμε βελτιώσεις ε, και στη συνεργασία που έχουμε με τα κράτη-μέλη για κάνουμε ιδιαίτερε προσπάθειε για τη σωστή αξιολόγηση τη πλεονάσια ικανότητα. Ε, Τέλο πάντων, εν ολίγη προσπαθούμε με κάθε μέσο να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση και να ε, προσεγγίσουμε στο μέτρο του δυνατού την κατάσταση όπω πραγματικά έχει για την πλεονάσια ικανότητα. Για τα θαλασσοπούλια τώρα, δεν είναι ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την έκθεση, αλλά ο κύριο Χάγκλου επέλεξε να συμπεριλάβει αυτό το θέμα ε, ασχολούμαστε και εμεί με τα θαλασσοπούλια, αλλά από μια κάπως διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση με τον κύριο Χάγκλουντ. Βάσει των αναλύσεων μας ε, μπορεί να επηρεάζονται τα θαλασσοπούλια όχι μόνο από τη θάλασσα και τα αποθέματα, αλλά και από την αλλιευτική δραστηριότητα και άρα η Επίτροπος ε, ε, δεσμεύτηκε για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για τα θαλασσοπούλια και την προστασία τους σε σχέση με τις ε, αλλιευτικές δραστηριότητες και προετοιμάζουμε ακόμη αυτό το σχέδιο δράσης. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχω δυστυχώς συγκεκριμένη ημερομηνία για την έγκριση, αλλά το επεξεργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο μένα, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα. Ε, άλλα δύο ζητήματα, ε, πρόσβαση στις, ε, στους πόρους και στην έκθεση και σε παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής. Προέκυψε ότι υπάρχει μια προτίμηση για μηχανισμούς που επιτρέπουν κατανομή αλλιευτικών ικανοτήτων και δικαιωμάτων επί τη βάση κάποιων κριτηρίων που σχετίζονται είτε με το χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ε, είτε με άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματο χάρη ε, οι κοινωνικές συνθήκες. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση. Το μόνο που είπαμε είναι ότι ουσιαστικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών για να προσδιορίσουμε ποιο τρόπο θα κατανείμουν τι ελευτικέ ικανότητε και τα ελευτικά δικαιώματα ανάμεσα στου αλληλεί και γι' αυτό το λόγο ε, απόσχομαι από τέτοιε συζητήσει. Η Επίτροπο όμω η ίδια σε μία ε, συνεδρία που έγινε εδώ στο Κοινοβούλιο ε, είπε ότι βρίσκει ιδιαίτερα ελκυστική την ιδέα αλλά δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει δικαιοδοσία. Τέλος, ένα τελευταίο σημείο που υπάρχει στην έκθεση είναι το Shetland Box. Δεν συζητήθηκε εδώ. Αληθεύει ε, ότι αυτό ε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του βασικού κανονισμού αυτή τη στιγμή, αλλά ε, προς το παρόν δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση για τον νέο βασικό κανονισμό. Να σας εξηγήσω ότι έχει γίνει ακόμη μία φορά, και μάλλον το ξέρετε, ε, αυτό το Shetland Box ε, ε, είναι ένας περιορισμός της αλλιευτικής δραστηριότητας σε βάση κριτηρίων που σχετίζονται με τη διατήρηση αποθεμάτων και όχι άλλων στοιχείων όπως η προστασία κάποιων στόλων ή κάποιων οικονομικών συμφερόντων των παρακτήων περιοχών. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια πολιτική διατήρηση, εργαλείο διατήρησης και άρα δεν πρέπει να ανήκει στο βασικό κανονισμό αλλά στα νέα τεχνικά μέτρα όπου θα ομαδοποιήσουμε όλα τα μέτρα διατήρησης αποθέματος που έχουν κάποια τεχνική πτυχή. Λοιπόν, γι' αυτό δεν τη συμπεριλάβαμε στη νέα πρόταση, γιατί θα συμπεριληφθεί στην πρόταση για τα νέα τεχνικά μέτρα ε, που θα καταθέσουμε αμέσω μετά την έγκριση του βασικού, ε, συγγνώμη, του βασικού κανονισμού και ε, αυτά προς το παρόν. Ο κύριος Ντέιβις θέλει να ρωτήσει κάτι την Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα αυτής της πλενώσης ικανότητα και των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη αναθεώρηση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Πολλοί αντιτίθενται στα TFC, παρότι μπορούν να χρησιμεύσουν για να μειώσουμε την πλεονάωσα ικανότητα. Προτείνεται μεταξύ άλλων να έχουμε τα TFC, εκτό και αν τα κράτη-μέλη βρουν κάποια εναλλακτική λύση για να μειώσουν την πλεονάωσα ικανότητα. Από ό,τι κατάλαβα και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου η κυρία Φράγα, οι επίτροπε είπε ότι θα καταθέσει προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ε, μέτρηση τη ικανότητα και άρα θα προκύψουν και εναλλακτικέ ε, λύσει ε, για να καταπολεμήσουν τα κράτη-μέλη αυτό το πρόβλημα. Δεν μου δώσατε την ίδια εντύπωση. Ε, ε, από ό,τι κατάλαβα, με έναν ασαφή τρόπο το μελετάτε ακόμη. Ε, και θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα, ε, πρωτού χρειάζεται να ψηφίσουμε για αυτό το θέμα. Ε, αναμένονται πρωτά, να περιμένουμε προτάσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ακριβείς. Το ήξερα ότι θα το θέσετε αυτό το ερώτημα. Δεν θα απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Η Επίτροπος θα έρθει εδώ σε 7-8 λεπτά. Εγώ δεν ε, θέλω να κάνω κάποια πρόταση, αλλά αν ε, ξέρετε τις ακριβείς ενδείξεις, εγώ δεν ήμουν εδώ όταν έλαβε χώρα η συνεδρία στην προηγούμενη φορά. Ε, εγώ όπως γνωρίζω δεν κάνουμε κάτι αόριστο μονίμως παρακολουθούμε την ικανότητα και μονίμως προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αξιολόγησή μας μαζί με τα κράτη-μέλη και είναι αρκετά δύσκολο να αξιολογήσουμε την κατάσταση του στόλου σε σχέση με την κατάσταση των αποθεμάτων και των πόρων. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που συνεχώς ε, μας απασχολεί, αλλά ε, τώρα δεν μπορώ να πω εδώ ξεκάθαρα ότι εκπονούμε έναν ορισμό για την πλειονότητα ικανότητα. Μαζί με το STCF ε, συνεργαζόμαστε στενά για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν έδω ορισμού, αλλά αν η Επιτροπή θέλει να σα αφήσει για την εκπόνηση αυτού του ορισμού, θα με ενδιαφέρει να το ακούσω κι εγώ. Δεν μπορώ λοιπόν να σα πω κάτι παραπάνω, πέρα από τι πληροφορίε που έχω εγώ στη διάθεσή μου. Μάλιστα, σα ευχαριστώ για να κλείσουμε τη συζήτηση. Κύριε Χάγκλουκ, το πολύ πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την πλεονάζουσα ικανότητα και την ανάγκη να έχουμε ορισμό. Και εγώ το συζήτησα το θέμα αυτό με την Επιτροπό και είχα πολύ μεγάλε ελπίδε ότι θα παρουσιάσει η Κομισιόν ένα σαφή ορισμό και μια εκτίμηση σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα για κάθε κράτο μέλο. Σε κάθε κράτο μέλο, αυτό είναι φυσικά κάτι που πρέπει να κάνουμε από κοινού. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό το έργο, στο να προσδιορίσουμε, να ορίσουμε την πλεονάζουσα ικανότητα γιατί αν δεν το πράξουμε, δεν είναι δυνατό για μας ε, να ζητήσουμε υποχρεωτικές με ελευτικές παραχωρήσεις. Αν δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε πώς ορίζουμε την πλονέσου ικανότητα, πώς μπορούμε να ζητήσουμε τι ευσύς. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου για τα καλά σχόλια. Θα τα λάβω υπόψη βεβαίω ε, σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κ. Μπεσέτ για τα TFC, τι μεταβάσει στι ελευθερικέ παραχωρήσει. Προσωπικά, εμένα δεν μου αρέσουν και τόσο, αλλά είδα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό με το πρόβλημα τη και ικανότητα σε ορισμένε περιοχέ ιδίω, γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε και αν δεν έχουμε άλλα εργαλεία να προτείνονται αξίζει να δοκιμάσουμε. λέγω προσωπικά είμαι ανοιχτό και σε άλλα μέτρα. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω. Για άλλε προτάσει, αν υπάρχουν, ευχαρίστω να τι υιοθετήσω. Και να συνεργαστούμε από αυτόν σε ό,τι αφορά το σχολείο του κ. Πυρίλο για την ισορροπία. Και σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λοβίν. Συμφωνώ, Ιζαμπέλα, με τον ορισμό σου αλλά εσύ έτσι ερμηνεύει την έκθεση. Το κύριο μήνυμα μου είναι ότι αν το χάρη, αν για οικολογικού λόγου, ε, ε, θέλουμε να περικόψουμε την ελευτική ικανότητα και τα, ποσά που, τα ποσοστά που αλλιεύονται πρέπει να έχουμε και κοινωνικά μέτρα να υποστηρίξουμε όσους οικονομικά θα φυγούν. Σε αυτό αναφέρομαι με την ισορροπία. Και φυσικά κάποιο μπορεί να ερμηνεύσει με πολλού τρόπου τον όρο ισορροπία. Εγώ κατάλαβα ότι διαφορετικά το κατάλαβε εσύ. Πρέπει να ξαναδούμε τη διατύπωση, τουλάχιστον για να συνεννοούμαστε για το σημείο αυτό. Φυσικά έχει δίκιο ότι χωρί οικολογική ισορροπία δεν θα έχουμε βιώσιμη ελεία οικονομικά στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ελεία μικρή κλίμακα, ελπίζω ότι μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να υποστηρίξουμε την αλία αυτή όσο είναι βιώσιμη, γιατί τώρα ως ένα βαθμό επιβάλλουμε τις ίδιες απαιτήσει και για την αλία μικρής κλίμακας, όπως ε, έχουμε και για την αλία μεγάλης κλίμακας. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο ή όχι, αλλά δεν θα μπω τώρα σε μεγάλη συζήτηση για το θέμα ε, για τις φώκες, αλλά μπορώ να σας δώσω αξιόπιστα στοιχεία για το μεγάλο αντίκτυπο που έχουν οι φώκες σε ορισμένες περιοχές. Και πράγματι ε, υπάρχει επίπτωση στην κατάσταση του χρειοποθέματος. Τώρα το, πρέπει να το βάλουμε αυτό εδώ σε αυτήν την εκθέση όχι. Δεν ε, ξέρω αν πρέπει να το συζητήσουμε εδώ, δεν θα συμφωνήσουμε ούτε για το κυνήγι της φώκιας. Εδώ, εμένα μπορεί να με ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα αυτό από κάποιο άλλο, αλλά υπάρχουν ε, ε, κάποια μέτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε τον αριθμό ε, των φωκιών, αλλά δεν θα τα συζητήσουμε εδώ αυτά. Πάντως σας ευχαριστώ όλους ε, για την ε, εξέβριση ενός καλού συμβιβασμού κατόπιν αυτών. Πρόεδρος Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 26 Μαρτίου επίσης. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών για να καλωσορίσουμε την κυρία Δεμανάκη όταν θα έρθει. Bueno, continuamos, si les parece. Damos la bienvenida a la Να συνεχίσουμε, να καλωσορίσουμε την κυρία Επίτροπο και χωρίς χρονομετριβή να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξη, το διαφρομένο διάλογο με την Επίτροπο Μαρία Δεμενάκη για τις πολιτικές και νομοθετικές προτεραιότητες για το 2013. Ξέρετε ότι έχουμε τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και όχι μόνο θα αξιολογήσουμε το πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2012, αλλά το σημαντικό είναι να προσδιοριστούν οι πολιτικές και νομοθετικές προτεραιότητες για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2013. Και στη βάση αυτή φυσικά θα ενημερώσω την Επιτροπή στην διάσκεψη των Προέδρων για τη σχετική συζήτηση. Βεβαίω θα υπάρχουν πάρα πολλέ προτάσεις και δεν ε, είμαι εγώ αρμόδιος να τα πω, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, είναι πολύ ξεκάθαρες ε, οι ιδέες και οι προτεραιότητες και ξέρετε πώς πρέπει να ε, περιορίσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το σύνολο, την μεγάλη βεντέλεια των θεμάτων ε, που έχει η Επιτροπή μας. Λοιπόν, για τη συζήτηση τώρα, καταρχήν θα λάβει το λόγο κυρία Επίτροπος ε, για 3-5 λεπτά και κατόπιν θα πάρουν το λόγο οι συντονιστές, περίπου 3-4 λεπτά ο καθένας και στη συνέχεια θα απαντήσει η κυρία Επίτροπος και τα τελευταία 20-25 λεπτά θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τους υπολείπους βουλευτές και θα απαντήσει η κυρία Επίτροπο στο τέλος. Έχουμε για όλα αυτά μία ώρα στη διάθεσή μας και εγώ όπως πάντα θέλω να σας ζητήσω να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι για να μπορέσουμε να έχουμε και χρόνο να ολοκληρώσουμε. Χωρίς χρονοτριβή έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές και αγαπητές, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα πάλι μαζί σας και να θα ακούσω τις προτεραιότητές σας για το χρόνο, για το, το χρόνο που μας μένει. Έχουμε το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Πριν ακούσω τις απόψεις σας, να πω λίγα λόγια για τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν νομίζω τους επόμενους μήνες. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη που θα πω ότι η έγκριση της μεταρρύθμισης είναι η πρώτη μας και πιο σημαντική προτεραιότητα. Όσο συντομότερα γίνει, εγκριθεί, εγκριθεί η μεταρρύθμιση, τόσο πιο γρήγορα θα επωφεληθεί ο κράτος. Να προχωρήσουμε δηλαδή προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης αλίας και να υποφεληθούν οι ψαράδες από περισσότερες δουλειές και έξτρα εισόδημα. Για να γίνει λειτουργική η μεταρρύθμιση θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να θεσπίσει guidelines, εφαρμοστικούς κανόνες και πρόσθετη νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις. Του χρόνου λοιπόν θα είναι το έτος που θα αφιερωθεί στην μεταρρύθμιση. Όταν θα τεθεί σε ισχύ ο βασικός κανονισμός θα χρειαστεί να αναπτύξουμε νέα σχέδια για την αλία βασισμένα σε πολιετή σχεδιασμό. Έχουμε κάποιες δυσκολίες για να προχωρήσουμε με αυτή την προσέγγιση και γνωρίζετε βεβαίως ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα μεταξύ ημών, του Κοινοβουλίου δηλαδή, και του Συμβουλίου Υπουργών. Του χρόνου θα πρέπει να υποβάλουμε επίσης τις πρώτες προτάσεις για να υλοποιηθεί η απαγόρευση απόρριψης στην θάλασσα και για τη δημιουργία του αλλιευτικού και θαλάσσιου ταμείου. Προς τα έξω θα διαπραγματευτούμε πρωτόκολλα και θα μεταμορφώσουμε τις συμφωνίες μας σε συμφωνίες βιώσιμης αλίας. Όλες οι νέες μας συμφωνίες θα ενταχθούν σε αυτή, θα εντάσσονται μάλλον σε αυτή τη νέα κατηγορία και θα περιλαμβάνουν ρήτρε διακυβέρνησης. Χθε το Συμβούλιο ενέκρινε τα πορίσματά του για την εξωτερική διάσταση της μεταρρύθμισης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη διότι είναι αυτό το πρώτο μέρος της μεταρρύθμισής μας που εγκρίνεται. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ώστε να επεκτείνουμε το ε, πεδίο ε, συμφωνιών μας και ιδίως για τον τόνο και με νέες χώρες. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους, ε, νέους, με τους διεθνείς εταίρους μας για τους ε, περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλίας, να ενισχύσουμε την επιστημονική βάση των οργανισμών αυτών και να αναλύσουμε τους λόγους της μη συμμόρφωσης και να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν το ιστορικό τους συμμόρφωσης. Φέτος θα γίνει η Ρίο και θα είναι βεβαίως ε, υψηλή προτεραιότητα, έχουμε ήδη προετοιμάσει τις θέσεις μας. Του χρόνου θα υποβάλω σχέδιο δράσεων Α, για τον Ατλαντικό ωκεανό. Και στην Κομισιόν επίσης προετοιμαζόμαστε για μια πολιτική για την Αρκτική, την οποία θα υποβάλουμε στις επόμενες εβδομάδες προσδοκώ την διαρκή σας συνεργασία για να αναπτύξουμε μια πολιτική η οποία θα είναι αυτάρκης και μια πολιτική η οποία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών μας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αναμένω λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ιδέες σας για το 2013. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αντινόρο καταρχήν έχει το λόγο από του συντονιστέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο και σας ευχαριστούμε γιατί για μια ακόμη φορά συναντιόμαστε στα πλαίσια λίγων εβδομάδων. Και εγώ θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις ε, για να καταλάβω αν μπορέσουμε να φτάσουμε και σε κάποια λύση για τα προβλήματα που έχουμε. Καταρχήν, ε, σε αυτό το έτος μία νέα πρόταση για τα τεχνικά μέτρα θα την έχουμε ή όχι, γιατί ξέρετε θα λήξει η παλιά πρόταση και κινδυνεύουμε ε, να έχουμε ένα νομοθετικό κενό στην επόμενη περίοδο. Και κατόπιν ε, για τα σχέδια ανασύσταση των πληθυσμών. Ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα διέξοδο, έχουν μπλοκαριστεί εργασίες μου φαίνεται ότι είναι παράλογο και δύο χρόνια μετά τι θέσει σε ισχύ τη Συνδική Λισαβόνα συνεχίζεται να μην γίνεται σεβαστή συναπόφαση σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ε, σε σχέση με αυτά τα σχέδια ανασύσταση του πληθυσμού και καλώ την κυρία Επίτροπα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να απεμπλοκαριστεί η κατάσταση αυτή να βγούμε από το αδιέξοδο κάτι ακόμα το οποίο το έχω πει και στο παρελθόν καθώς ε, ε, στο εσωτερικό της ε, ομάδας μας έχουμε διάφορες όμορες χώρες που αλλιεύουν ε, και το πρόβλημα είναι να κατορθώσουμε να ρυθμίσουμε τη σχέση με τις όμορες χώρες. Δηλαδή εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε στους, ε, να επιβάλλουμε κανόνες στους δικούς μας αλληλείς και οι άλλοι συνεχίζουν να μην ε, υποβάλλονται στους ίδιους κανόνες και συνεχίζουμε δηλαδή να επιβάλλουμε κανόνες στην Ευρώπη και τελικά οι άλλοι κατορθώνουν να συνεχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν θα μπορέσουμε τελικά να συμφωνήσουμε με αυτές τις όμορες χώρες για να μπορέσουμε όλοι μας να ρυθμίσουμε την, την αλία. Και κατόπιν για τις ε, βιώσιμες συμφωνίες αλίας, έτσι όπως ε, ορίστηκαν από εσά με το νέο κανόνα. Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη, έχουν υποθεί κάποια, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία από τώρα για να μπορέσουμε να διαρθρώσουμε καλύτερα τη συζήτηση για το μέλλον ευχαριστώ. κύριε Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που είστε πάλι κοντά μας σήμερα και θα ήθελα να έρθω στα γενικά πρώτα της γενικής αλληλευτικής πολιτικής. Πιστεύω ότι η ισχύουσα κοινή αλληλευτική πολιτική έχει αποτύχει έχει αποδειχθεί ότι τα σημαντικά προβλήματα όπως της υπεραλίευσης, της υπερβολικής χωρητικότητας των σκαφών, της κακής κατάστασης του αλληλευτικού τομέα, τα κοινωνικά προβλήματα κλπ. λόγω της μείωσης των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων σε πολλές ε, παράκτητες περιοχές έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντικά προβλήματα. Κυρία Επίτροπε, έχετε υποβάλει σχέδια για μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση. Η πολιτική μας ομάδα σας εγγυώμαι ότι θα συνεργαστεί μαζί σας με την ελπίδα να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα. Με την έννοια αυτή είναι σημαντικό για μας να σημειώσουμε ότι η κατάσταση στη Μεσόγειο διαφέρει από άλλες θάλασσες που βρέχουν την Ευρώπη. Τα, τα ε, αλληλευτικά αποθέματα έχουν εξαντληθεί, είναι λίγα και τα μοιράζονται πολλές χώρες μέλη το ερώτημά μου είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η πρότασή μας είναι χρειαζόμαστε μια προσαρμοσμένη κοινή αλληλευτική πολιτική και για την Μεσόγειο. Χρειαζόμαστε και εκεί μια μεταρρύθμιση. Τι θα κάνουμε, ποιες ιδέες έχετε εν προκειμένου. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα με τη διαδικασία συναποφάσεως. Δεν μας φαίνεται ρεαλιστικό η θέση σε ισχύ του νομοθετικού πακέτου να γινει πρώτη πρώτου του 2013. Εν προκειμένου θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεωρήσει τις δύο νομοθετικές προτάσεις ως κατεπίγουσες και να τους δώσει την ύψιστη δυνατή προτεραιότητα. Έρχομαι και στο άρθρο 17.2 Γενική όρη πρόσβασης και περιορισμοί ο βασικός κανονισμός που ισχύει τώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι ότου εκδοθεί νέος, έτσι υποθέτω, με εξαίρεση μιας ρήτρα του άρθρου 17 παράγραφος 2 για την πρόσβαση περιορισμών σε 12 μίλια που λύγει τώρα μέσα στο 2012. Εάν εγκριθεί νέος κανονισμός, τότε οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θα ισχύουν πλέον. Για να αποφευθεί αυτό, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει προτάσεις για, που να προβλέπουν παράταση της ισχύω των διατάξεων του άρθρου αυτού, ώστε να μπορέσει να περιληφθεί στην νομοθετική διαδικασία. Έχω ακόμα λίγες ερωτήσεις, αλλά θα αρκεστώ για την ώρα σε αυτές για να μην υπερβώ το χρόνο. Γκάλαχερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε σήμερα το απόγευμα για να συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασίας για τους επόμενους μήνες και φυσικά το επόμενο έτος. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα που δεν αναφέρθηκαν και που με απασχολούν. Ποια πρόοδο προσδοκάτε σε σχέση ε, με την προσωρινή κατάσταση και την αποτελμάτωση που υπάρχει, δηλαδή 43-2 και 43-3 στη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι ένα διέξοδο διότι ε, αποφασίζουμε για ζητήματα ζητήματα βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα που μα απασχολήσουν σε δύο ή τρία χρόνια. Όμω δεν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα στα προβλήματα που άμεσα μπορούμε να ρυθμίσουμε, διότι είναι ντροπή. Από την 1η Δεκεμβρίου του 2009 έχουμε σημειώσει μηδενική πρόοδο για κάποια ζητήματα, ενώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει, παραδείγματο χάρη, ε, μακροπρόθεσμη διαχείριση για τον βορείο Ανατολικό Ατλαντικό για το ε, σκουμπρί. Για το σαφρίδι, συγγνώμη. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να έρθει νέα εντολή, νέα επιτροπή, νέα επίτροπος. Είναι ως επίτροπος, μα δεν είναι λύση. Αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, και να κινηθούμε, διότι πώς θα εξηγήσουμε στο κοινό. Δηλαδή, τι θα σκεφτούν, στέλνουμε αυτού στο κοινοβούλιο και δεν μπορούν να λύσουν ένα τόσο απλό ζήτημα και ασχολούμαστε με τον έλεγχο των αλλιευμάτων και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ε, να αυτά τα βασικά ζητήματα. Ε, ε, δεν μπορείτε, ε, εν πάση περιπτώσει, να βρείτε μία λύση. Πάντοτε συμβαίνει αυτό, δηλαδή ε, ε, ε, συζητούμε για δυσεπίλητα ζητήματα ενώ δεν ρυθμίζουμε τα άμεσα αυτά που είναι εύκολο να ρυθμίσουμε μπορείτε να προτείνετε και να κάνετε κάτι σε σχέση τώρα με το πλαίσιο των τεχνικών μέτρων ξέρουμε ότι τα ε, τεχνικά μέτρα ο κανονισμός των τεχνικών μέτρων θα εκπνεύσει στα τέλη του 2012 και ξέρω ότι δεν είστε από αυτούς που θα μετακύλιαν θα παρέτειναν την ισχύ του ζητήματος εγώ προτείνω το ταχύτερο δυνατόν να επανέλθετε και να προτείνετε τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση μετά το 2012 ως προς τις εμπορικές κυρώσεις τις ε, πραγματευόμαστε εδώ, αλλά χρειαζόμαστε ένα νέο στοιχείο. Πρέπει να ρυθμίσουμε την κατάσταση και πάλι δεν ξέρω, αλλά ε, ε, και υποθέτω ότι είναι μεγάλο το άχθος που σας βαραίνει. Όμως η υπηρεσία σας δεν θα έπρεπε επιτέλους ε, να ε, βρουν ένα πρόβλημα αυτών των τεσσάρων κρατών μελών ε, που συνιστούν εμπόδιο. Μπορούμε να έχουμε τις κυρώσεις, δεν χρειάζεται να τις εφαρμόσουμε, αλλά να υπάρχει το πλαίσιο, δηλαδή να έχουμε αυτό το απαραίτητο εργαλείο θα προτιμούσα, όλοι θα προτιμούσαν να συνεργαστούν αυτά τα τέσσερα κράτη. Αν τα αφήσουμε μέχρι το τέλος του έτους, ξέρετε, θα συμβεί για το 2013 θα έχουμε μία μια μονομερή δήλωση και θα συνεχιστεί όσο έχει η κατάσταση ε, επί σειρά ετών και αυτό εξισούται με καταστροφή ε, του κλάδου. Ε, γι' αυτό και σε αυτό το στάδιο σας επισημαίνουμε αυτά τα ζητήματα. Φυσικά επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για το μέλλον αν δεν λύνουμε τα προβλήματα του παρόντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κάλλη και κυρία Λεβέντη. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Φυσικά οι προσδοκίες από το 2013 θα είναι να έχουμε το νέο βασικό κανονισμό και να ισχύει και η νέα κοινή ελευτική πολιτική. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο έργο για το μέλλον, όμως αν πρέπει να θέσουμε κάποια προτεραιότητα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η απαγόρευση απορρίψεων οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των περιπτώτων των ελευμάτων. Δεν ε, θα είναι λοιπόν μόνο υποχρέωση εκφόρτωση των πάντων, αλλά πράγματι θα μειώσει τα περιπτώντα ελεύματα. Αυτό που πρέπει να είναι ο στόχο τη απαγόρευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πλειονότητα ικανότητα. Αν ε, δεν υπάρχει σύστημα μεταβάσιμων ελευτικών παραχωρήσεων που να λειτουργεί, τι θα κάνουμε με αυτή την πλεονάζουσα ικανότητα, πώ θα τη διαχειριστούμε. Τέθηκαν ε, αρκετές ερωτήσεις αυτή την Επιτροπή σήμερα για τον ορισμό της πλεονάζουσας ικανότητας. Πρέπει να παρακολουθούμε τα κράτη-μέλη και προκειμένου να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός της πλεονάζουσας ικανότητας και κάποια παρακολούθηση της μείωσης της πραγματικής πλεονάζουσας ικανότητας. Θα ήθελα κάποια σχόλια από αυτού. Τώρα, για την εξωτερική διάσταση, νομίζω ότι η διαφάνεια για τις αλευτικές συμφωνίες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα ήταν ε, πολύ καλό να γίνει μια πολύ καλή δουλειά στη διαπραγμάτευση με τις τρίτες χώρες, δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σε όλη την ελευτική πίεση σε αυτά τα ύδατα, για να είμαστε σίγουροι ότι διαπραγματευόμαστε μόνο επί του πλεονάσματος, του αποθέματος, το οποίο δεν χρειάζεται η χώρα αυτή, και για την αλλή απλά ε, θα ήθελα η Κομισιόν ε, να προχωρήσει με την έκθεση που θετήθηκε από το Κοινοβούλιο για το σύστημα ε, τεκμηρίωσης ελευμάτων. Θέλω, θα, ξέρω ότι θέλει να το κάνει η Κομισιόν και είναι προτεραιότητα και πρέπει και να το βελτιώσουμε γιατί χρειαζόμαστε πραγματική χνηλσιμότητα και όχι απλώς χαρτιά. Ξέρουμε ότι όλα τα ψάρια που τίθενται σε εμπορία παγκοσμίω πρέπει να προέρχονται από, βιώσιμε πηγέ και για το Ρίο Συνικό. Συγχαίρω την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πολύ ε, υψηλά στην ατζέντα του ωκεανού. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε και όσα συμφωνήθηκαν στο Ρίο και χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό συντονιστικό στο υψηλότερο επίπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο ε, στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση των ωκεανών. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να το προωθήσουμε αυτό και ε, στην συνάντηση Ρίο 20 θα είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Αυτές είναι οι προτεραιότητες λοιπόν από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβενσον. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο που είναι παρούσα εδώ. Αύριο, εδώ, αύριο το απόγευμα, διεξάγεται ακρόαση για την περιφερειοποίηση και θα μας διευκολύνετε αν μας πείτε, κύριε Επίτροπε, ότι συμφωνείτε με τη διαχείριση των χωρών μελών και ότι η Κομισιόν θα διατηρήσει το δικαίωμα να καθορίζει το πλαίσιο και θα ανακαλέσει στη τάξη κάθε χώρα η οποία δεν θα συμμορφωθεί. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και για τη μικροδιαχείριση που και εσείς επικρίνετε. Το θέμα των απορρίψεων στο, στο χθεσινό συμβούλιο, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν κατατέθηκε τροπολογία από χώρες μέλη που είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι οι τροπολογίες για να αποδυναμωθεί η απαγόρευση των απορρίψεων. Σας ρωτώ όμως εάν συμφωνείτε με την αντίληψη της κυρίας Ροντούστ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ανά είδος αλίας και όχι ανά είδος ψαριού και να είναι μια προσέγγιση και κινήτρων και αντικινήτρων και, και μαστιγιού και καρότου δηλαδή και με τεχνικά μέτρα δίνοντάς τους έξτρα μέρες στη θάλασσα ή έξτρα ποσοστώσεις, αλλά και με επιβολή κυρώσεων. Και όπως προτείνει η κυρία Ροντούστ, όταν θα φέρουν στις σκάλες νεαρά ψάρια, να τους μειώνουν οι ποσοστώσεις. Να επιβάλλονται δηλαδή έξτρα κυρώσεις Αυτές νομίζω είναι κάποιε καινοτόμε ιδέες της κυρία Ροντούστ. Και από ό,τι μαθαίνω ορισμένε συζητήθηκαν χθε στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις από αυτόν. Ευχαριστώ κύριο Φερέιρα. Τελευταίος από τους συντονιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσίαση. Θέλω να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Ε, το ένα το ακούσαμε ήδη από τη συνάδελφο Ρόντουστ και σχετίζεται με την καθυστέρηση την προβλεπόμενη καθυστέρηση ε, σε σχέση με τις ε, προτάσεις της μεταρρύθμισης. Και η συγκεκριμένη πρόταση που έχουμε, όπως είπε και η κυρία Ρόντουστ, ή μάλλον η μία ανησυχία που έχουμε σχετίζεται με το 17 β για την πρόσβαση στα ύδατα και τον ε, περιορισμό της ε, πρόσβασης που σχετίζεται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη των 12 μιλίων. Ε, υπάρχει κάποιος λόγος που αντιμετωπίζουμε αυτό το νομικό κενό ή χειρότερα ακόμη ε, μπορούμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τις προθεσμίες που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση της παράτασης αυτού του καθεστώτος ε, μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου βασικού κανονισμού. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη, ε, σχετίζεται με την ε, παράκτη αεραστεχνική αλία μικρής κλίμακας. Ε, η Επιτροπή γνωρίζει ήδη κατά πάσα πιθανότητα ότι το Κοινοβούλιο προτίθεται να συντάξει έκθεση πρωτοβουλία για την αλία μικρή κλίμακα και σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση κοινή αλλιευτική πολιτική μεταξύ άλλων για να καταδείξει ότι αυτό το τμήμα του κλάδου δεν έχει ε, εξεταστεί επαρκώς ε, ε, μέσα στι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, κάποιες προτάσεις μεταξύ άλλων και νομοθετικές ε, που αποσκοπούν στην παρέμβαση για να ρυθμιστούν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα της ε, αλίας μικρής κλίμακας υπάρχουν, υπάρχουν σχετικές ε, προθέσεις ε, για τις νομοθετικές προτάσεις σας το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να λάβει υπόψη τις ιδέες που ενδεχομένως να ανακύψουν για αυτό το θέμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα παρουσιαστούν υπό τη μορφή, όπως σας είπα, μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβούλια. Ε, θα ήθελα να εξασφαλίσω από πλευρά σα ότι προτίθεστε να τι λάβετε υπόψη για να καλύψουμε τι εφιστάμενες ατέλειες ε, των γνωστών προτάσεων, είτε σχετίζονται με τον βασικό κανονισμό, είτε με την κοινή οργάνωση αγορά, είτε με το ε, αλληλευτικό και θαλάσσιο ταμείο. Μία άλλη ερώτηση τώρα που έχετε ξανακούσει ε, φυσικά σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων και την υποχρέωση των κρατών μελών για την προσκόμιση δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση των αποθεμάτων. Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ε, την ε, ε, την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά όριο σε ποσοστό 50%. Και ρωτώ, στις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδώσει το απαιτούμενο βάρος σε αυτό το θέμα και στο μέλλον πάλι για τη συλλογή των δεδομένων ποιες είναι οι προθέσεις σας. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωση, ούτω ώστε να υπερβεί αυτό το 50% που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία όπως σα έλεγα ω ανώτατο όριο. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερέιρα. Ε, θα ακούσουμε τώρα την Επίτροπο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις σε σχέση με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης, αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, ε, ε, οποιαδήποτε προτεραιότητα σχετίζουμε με τη μεταρρύθμιση σχετίζεται και με την πολιτική και με τους πόρους. Όταν δεν έχουμε επαρκείς πόρους, ε, φυσικά θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό και θα σε εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται ούτω ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το νομικό κενό. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα προκύψει αυτό το νομικό κενό. Ήδη έχουμε εξετάσει την κατάσταση, είμαστε έτοιμοι ακόμη και για το καθεστώ των 12 μιλίων. Δεν θέλουμε να το τροποποιήσουμε, θα προτείνουμε επιμήκυνση και για τα τεχνικά μέτρα ε, κάνουμε όλε τι απαιτούμενε προετοιμασίε. Μην ανησυχείτε, νομικό κενό δεν θα υπάρξει. Αλλά θέλω να σα πω, ε, να εκφράσω τη δική μου άποψη, ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να επισπεύσουμε τι εργασίε μα εν ώψη της μεταρρύθμισης, ώστε να έχουμε στα ε, χέρια μας σύντομα τον ε, νέο βασικό κανονισμό τους, ώστε να εγκριθεί γέρος. Για τη Μεσόγειο, ε, ακούσαμε δύο παρεμβάσεις, κυρίας το και του κυρίου Αντινόρη. Θα απαντήσω ως εξή. Ναι, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να ισχύουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπως είπε ο κύριος Σαντινόρη, και όντως έχουμε πολλά προβλήματα με τις γειτονικέ χώρες. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη περίοδο και στη Γενική Αλληλευτική Επιτροπή για την ε, Μεσόγειο, που είναι η αρμόδια επιτροπή για τη συνεργασία των ε, χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου. Τον συνάντησα στη Ρώμη, Ιταλός ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ε, επανειλημμένα έχω πάει στην έδρα αυτή της Επιτροπής και πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο συζήτηση για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά, θα είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει. Πάντω ευελπιστώ ότι κατά τι θα βελτιώσουμε την κατάσταση για την ε, μεταρρύθμιση. Χτε ε, το Συμβούλιο και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη συνεδρίαση στο Συμβούλιο. Συζητήσαμε και αυτό το θέμα, μεταξύ άλλων το θέμα της Μεσογείου και πρότεινα εγώ να έχουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για την ε, Μεσόγειο αναφερόμενη όλος ιδιαίτερο στη μεικτή αλία και τα προβλήματα ε, της μικτής αλίας ε, στη Μεσόγειο που σχετίζονται με τις απορρίψεις και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. συζήτησα αυτά τα θέματα επίσης με τους υπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας και εν ολίγης θεωρώ ότι πρέπει να προκρίνουμε αυτή την προσέγγιση αλλά θα πρέπει να, οι κανόνες που ισχύουν γενικότερα στη μεταρρύθμιση να ισχύουν και για την Μεσόγειο. Αυτό το ξεκαθάρισε ε, αποτινόμενη προς ε, όλες τις κυβερνήσεις και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό που δεν υπήρξε μονομερής ε, δήλωση κύριε Στίβενσον ε, ούτε καμία μονομερής πρόταση δεν προέκυψε τίποτα μίλησα ευθέω. χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση και για τη Μεσόγειο ναι χρειαζόμαστε ειδικέ λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες για κάποια ζητήματα αλλά δεν γίνεται να αποκλείσουμε τη Μεσόγειο από την μεταρρύθμιση ρύθμιση διότι αυτό δεν συνιστά τη θέμένη αξία και ούτε πρόκειται να το δεχτούν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Για να είμαι ειλικρινή μα, δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική τη συμμόρφωση, το καθεστώ μόνο για τι βόρειε χώρε. Ας θυμηθούμε επίσης ότι η υπεραλίευση ανέρχεται στο 80% στη Μεσόγειο, ενώ στη Βόρειο Θάλασσα δεν υπερβαίνει το 50%. Αυτό το χάσμα πρέπει να το καλύψουμε. Συζητήσαμε όμως κάποιες ειδικέ λύσεις. Αναφέρομαι και σε μία πρόταση του κυρίου, του κυρίου Μιλάνα. Πού είστε? Εδώ είστε. Ε, ο κύριο Μιλάνα ε, πρότεινε την δυνατότητα αποκλεισμού κάποιων ε, περιοχών για να προστατεύσουμε τους γεννήτορε, για την αναπαραγωγή δηλαδή και κάποια άλλα προβλήματα όπως παραδείγματο χάρη η κατανάλωση των νυχθιδίων στη Μεσόγειο. Οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε μια λύση γι' αυτό και η κυρία ρόντου θα έχει κάποιε προτάσει. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση με τον Ιταλό Υπουργό Αλία και ελπίζω ότι το Μάιο που θα ξανασυζητήσουμε την απαγόρευση ή των απορρίψεων θα έχει το Συμβούλιο πιο συγκεκριμένε προτάσει για την Μεσόγειο. Οπότε για τη Μεσόγειο ειδικέ λύσει, ειδικά προσαρμογέ, ναι, αλλά μέσα στο πλαίσιο τη συνολικότερη μεταρρύθμιση και ε, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη ε, το έχουν ε, δεχτεί και είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Πιστεύω ότι η πιο σημαντική απόφαση που ελήφθη χθε στο Συμβούλιο σχετιζόταν με την απαγόρευση των απορρίψεων, ότι αποφασίστηκε λοιπόν ότι Υποστηρίζουμε την καταληκτική ημερομηνία για την αρχή να ισχύει η απαγόρευση. Είχα επιμείνει όλο ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Επεξή, θα συζητάει το Συμβούλιο τον τρόπο με τον οποίο ε, θα επιτευχθεί ο στόχο και όχι το αν θα τεθεί αυτό ο στόχο τη απαγόρευση. Πώ, όχι αν. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το στοιχείο. Καλωσορίζω την πρόταση. Ε, υπενθυμίζω ότι η Δανική Προεδρία μας βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολύ το τονίζω, ε, για την εξέβρεση της λύσης. Ε, επίσης, ε, προτείνω από κοινού με τη Δανική Προεδρία και βάσει μιας ιδέας ε, που είχε ε, εισηγηθεί η κυρία Ρόντου στο ότι θα βασιζόμαστε στα αλλιεύματα και όχι στα είδη. Ναι, θα αποφασίσουμε για την απαγόρευση επί τη βάση των αλλιευμάτων και όχι των ειδών. Το αποφάσισε ήδη αυτό το Συμβούλιο ε, και είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας για να βρούμε λύσεις. Αν αλλιεύμα λοιπόν θα αποφασίζεται η απαγόρευση, σταδιακή προσέγγιση φυσικά, καταληκτική ημερομηνία, θα δούμε πότε θα είναι αυτή. και ελπίζω ότι ε, δεν θα γίνουν άλλες συζητήσεις σχετικά με το αν θα επιβληθεί αυτή η απαγόρευση. Θα συζητάμε μόνο τον τρόπο, τα προβλήματα εφαρμογής, τα πρακτικά προβλήματα κυρίως για τη μεικτή ε, για τα μεικτά αλλιεύματα και τα ε, μέτρα που πρέπει να λάβουμε άμεσα. Πάλι σε σχέση με την απαγόρευση των απορρίψεων, θα ήθελα να επαναλάβω, απαντώντας και στην κυρία Λεβίν, προσπάθησα να το εξηγήσω νωρίτερα, λοιπόν, ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν είναι απροετοίμαστη να πάει ε, στην απαγόρευση. Η επιλεκτικότητα του εξοπλισμού είναι πρωταρχική ε, σημασίας. Θέλουμε νέες ιδέες για νέους εξοπλισμούς, ώστε να επιτύχουμε αυξημένη επιλεξιμότητα Ε, και αν ε, το επιτύχουμε αυτό θα είναι υψηλότερο το ποσοστό της συγχρηματοδότησης. Ε, η ΣΤΕΦΚ επίσης θα μας δώσει ένα κατάλογο ειδών με υψηλά ποσοστά επιβίωσης για να αποκλειστούν από τον κατάλογο του, της απαγόρευσης των απορρίψεων. Πολύ θετικά αυτά σε σχέση με τα ηχθίδια δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τους προσεχείς μήνες θα γίνουν πολλές τεχνικές συνεδριάσεις. Θα ξανασυζητήσουμε το Μάιο την απαγόρευση απορρίψεων και μέχρι τότε ελπίζω ότι θα έχει υποβάλει και το Κοινοβούλιο Τροπολογής για να μας δώσει ιδέες. Ε, όπως βλέπετε πάντως χρησιμοποιούμε ε, ε, ε, στο έπακρον της προτάσεις μη διστάζετε να υποβάλλετε τροπολογίες. Ως προς τα εμπορικά μέτρα και αυτό το νέο εργαλείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γκάλαχερ. Λοιπόν, αυτό το νέο εργαλείο είναι το καλύτερο που μπορέσαμε να πετύχουμε βάσει των νομικών συμβουλών που είχαμε στη διάθεσή μας. Αντιλαμβάνουμε ότι έχετε κάποιες προτάσεις Υπάρχουν προτάσεις για να διευρύνουμε το πλαίσιο και τη χρήση αυτού του νέου εργαλείου. Θέλω να εξετάσω αυτές τις προτάσεις για να δω αν υπάρχει ένα ε, περιθώριο ελιγμών, αν υπάρχει ένας νομικός τρόπος ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο εργαλείο. Στα παρασκήνια του Συμβουλίου επίσης κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για αυτό το πρόβλημα ε, της Ισλανδίας και των Ίσων Φαρόε δηλαδή, ας το πούμε, και για τις ε, παράκτες συμφωνίες τη Συμφωνία των Παράκτων Κρατών μάλλον. Ε, όλοι θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την επόμενη ημέρα. Θα χάσουμε άλλη, άλλη μία χρονιά ενώ είναι σε ε, ιδιαίτερα επισφαλή θέση το απόθεμα. Δεν ε, μας παίρνει αν θέλετε να χάσουμε άλλον ένα χρόνο και ζητώ επίσπευση των εργασιών από πλευρά ε, του Κοινοβουλίου στο μέτρο του δυνατού εξυπακούεται. Ε, το Συμβούλιο αποφάσισε να κινηθεί το ταχύτερο δυνατόν ούτω ώστε να τεθεί σε ισχύ ε, αυτό το νέο μέσο ταχύτερο δυνατόν. Ω προ το θεσμικό πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκατε ε, πολύ, δηλαδή η διαφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με την εφαρμογή ε, των άρθρων τη συνθήκη, τα ζητήματα τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και άλλα συναφή. Λοιπόν, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνω τη συζήτηση. Δεν αγνοούμε το πρόβλημα αλλά οφείλω να πω ότι είμαι μάλλον απογοητευμένη, ε, διότι βλέπω ότι δεν υπάρχει διαλλακτικότητα ε, στις διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ πεισματάρικα, δεν ε, υπάρχει κανένα περιθώριο ελιγμών και προσπαθούμε και ξανά προσπαθούμε με τους τριμερείς διαλόγους να βρούμε μία λύση αλλά νομίζω ότι ε, εκφεύγει των προσωπικών μου ορίων και της αρμοδιότητάς μου. Αν έχετε εσείς ε, κάποιες νέες ιδέες ε, παρακαλώ αλλά ε, Όντω ε, πρόκειται για ένα τέλμα και είναι ένα θέμα ε, θεσμικό ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να σας βοηθήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση για την πλεονάζουσα ικανότητα και εν γέννη τα προβλήματα της αλληλευτικής ικανότητα. Ξέρω ότι ε, υπάρχει διάσταση απόψεων σε σχέση με τον ορισμό της ε, αλληλευτικής ικανότητα, τη πλεονάζουσα ικανότητα κτλ. Λοιπόν, αποφάσισα ε, του επόμενου μήνε να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα θέμα που είναι σαφέστατο, ελέγξιμο και τα κράτη-μέλη έχουν την απέτηση να υποβάλουν εκθέσεις στην γενική μα διεύθυνση μέχρι το τέλο του έτου. Η ισχύ των κινητήρων, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή αναμένεται εθνική ετήσια έκθεση μέχρι το τέλος ε, του 2012 ε, για αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο ε, και στο παρελθόν έχουν γίνει πολλά, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Πάντως τα δεδομένα που πήρα εγώ στα χέρια μου όταν ανέλαβα είναι τουλάχιστον ανεπαρκεία, το θέσω έτσι. τώρα θα τους υποχρεώσω πολύ συγκεκριμένα να κάνουμε μια αξιολόγηση της ε, κατάστασης. Ε, πρόκειται για, ένα, ε, για πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και θα ήθελα να λάβουμε αυτές τις εκθέσεις και παρακαλώ όποιος έχει προτάσεις να μην διστάσει. Πάντως έχω συζητήσει με αυτά τα κράτη-μέλη και δεν έχουμε προς το παρόν αρκετά καλές προτάσεις, οπότε θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα τον Απρίλιο στην επόμενη σύσκεψη του Συμβουλίου για τις ε, μεταβάσιμες ε, παραχωρήσεις ε, και ελπίζω να, να, έχω μια πρώτη εικόνα για την ισχύ των κινητήρων. Μόνο τρία κράτη-μέλη προς το παρόν έχουν δώσει στοιχεία, ούτω ώστε να περιγράφουν επαρκώς την, την κατάσταση στη χώρα τους για αυτό το ζήτημα και αντλούμε πάρα πολλέ πληροφορίες από αυτά τα στοιχεία που μα δίνουν. ω προς την εξωτερική διάσταση τώρα, της ε, κοινής αλλιευτικής ε, πολιτικής ε, έχουμε νέο κεφάλαιο αυτού στην προτινόμενη μεταρρύθμιση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εγκρίθηκαν ήδη, όπως σας είπα, για την εξωτερική διάσταση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής και τα συμπεράσματα αυτά συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά που προτείνεται και θα ήθελα να ε, επικροτήσω και πάλι το έργο της Δανικής ε, Προεδρίας. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα η πρότασή μας για τον νέο κανονισμό θα πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο πλαίσιο. Εφόσον ελήφθη αυτή η απόφαση από το Συμβούλιο πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτήν. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμη σκληρότερα για τα FPAs. Ε, για τις ε, αλλιευτικές ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Δηλαδή, συμφωνούμε για τη διαφάνεια, για όλες τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσουμε, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε σε κάποιο βαθμό. αλλιώ. Ε, Αυτό ελοχεύει ο κίνδυνο απώλειας όλων των συμφωνιών ε, και οι άλλε χώρες ε, θα έρθουν και θα πάρουν όλες τις αλληλευτικέ ικανότητε. Στο Μαρόκο, στη Μαυρετανία, το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Προσπαθούμε να βρούμε νέους εταίρους. Έχουμε τις Σεϊχέλες, το Μαυρίκιο, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι αρκετά μεγάλες συμφωνίες τους ώστε να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η Μαυριτανία. Ε, πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Αλλιώς ας προετοιμαστούμε όλοι για το ενδεχόμενο ότι θα χάσουμε αυτή την ε, δυνατότητα που έχουμε και δεν νομίζω να είναι θετικό για κανέναν, ούτε για τον κλάδο μας, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την ε, διαφάνεια, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και για τις ίδιες τις χώρες. Ε, φαντά, καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη διαφάνειας και όλα τα τα υπόλοιπα ε, ζητήματα είναι πάρα πολύ καλά για τις κυβερνήσεις αλλά για τους λαούς των χωρών αυτών σίγουρα δεν είναι καλές. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Για την περιφερειοποίηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, και αυτό θα το συζητήσουμε στην επόμενη σύσκεψη του Συμβουλίου ε, και ελπίζω να ακουστούν καινούργιες ιδέες ε, και ελπίζω να μας βοηθήσετε για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς αυτή την άσκηση. Για τα μικρά σκάφη και την ε, αλία μικρής κλίμακας προτείνουμε να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότηση και να φτάσει μέχρι και 75% ε, στα πλαίσια της νέας αλλιευτική πολιτική. Προτείνουμε να εξετάσω όλε τι δυνατότητε που υπάρχουν για να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα μικρά σκάφη. Θα εξετάσω τις προτάσεις και τις εκθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Πέντε. Δύο λεπτά ο καθένας για να υπάρχει και χρόνος για την απάντηση. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βαλέσα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Κομισιόν ε, προετοιμάζει την εισαγωγή πολλών σχεδίων ε, διαχείρισης αποθεμάτων ε, κυρίως για το γάδο και για τα πελαγικά είδη στη Βαλτική. επιστημονική κοινότητα και οι αλείς μας λένε σήμερα ότι το απόθεμα του γάδου τα πάει πολύ καλά, είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι πολύ θετικό για τους αλείς, αλλά υπάρχει απειλή για τα αποθέματα ρέγκας και σαρδελόρεγκας. Υπάρχει στην ε, Βαλτική ε, ένα ζήτημα ε, με αυτά τα αποθέματα και πρέπει να μπορέσουμε να επιτρέψουμε και την ανασύσταση του αποθέματος σαρδελόρεγκας αυξάνοντας την ποσόστοση για το γάδο. Έτσι λοιπόν στο μέλλον μπορεί να δούμε μείωση του σπράτ στη Βαλτική και πώς ε, μπορούμε να έχουμε μία πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση από την Κομισιόν. Μήπως η Κομισιόν σκέφτεται ότι τα σχέδια διαχείρισης ε, ε, θα έπρεπε να είναι ευέλικτα για να μπορούν να προσαρμόζονται στο επίπεδο του αποθέματος βάση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Μήπως θα έπρεπε να προβλέψουμε ένα περιθώριο λιγμών μεγαλύτερο για να μπορέσουμε να προσαρμοζόμαστε στο επίπεδο ε, του αποθέματος και στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, το Συμβούλιο πήρε κάποιες φιλόδοξες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα τάξη στη Βαλτική. Και προφανώ, αυτό ήταν απαραίτητο από βιολογική σκοπιά, αλλά οι συνέπειε ήταν ιδιαίτερα αρνητικέ. Ε, αναφέρομαι στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που υπήρξαν στους στόλους των χωρών της Βαλτικής. Πρόκειται για τη μείωση των τάκ και τα πελαγικά είδη. Αυτά τα τάκ ε, μειώθηκαν ε, λόγω ε, αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών που η Δήμη πως φέτος η Κομισιόν θα δείξει μεγαλύτερη κατανόηση για τους τόλους της Βαλτικής, λαμβάνοντα υπόψη και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Μία για το Μαρόκο εγώ θα είμαι συγγήτρια για την συμφωνία με το Μαρόκο από την πλευρά του Κοινοβουλίου και είμαι δετεθμένη να συνεργαστούμε πλήρως ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα μέσω του δυνατόν καλύτερο τρόπο. Ξέρω ότι στι 20 του μήνα εσεί ε, θα μεταβείτε στο Μαρόκο, οπότε υπολογίζετε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, στο καλύτερο δυνατό πνεύμα. Και δεύτερον, θα ήθελα να μιλήσω για κάτι που αναφέρατε εσείς ε, στη συνεδρίαση του ΕΛΚ της προάλλες σε σχέση με μια μελέτη για την πλεονέσουσα ικανότητα που υλοποιεί η Κομισιόν. Νομίζω ότι το αναφέρατε, αλλά δεν ήταν αρκετά σαφές. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της μελέτης και θα καθορίσετε απλώς κάποιες παραμέτρους και κατόπιν θα είναι τα κράτη-μέλη αυτά που θα αξιολογήσουν το θέμα αυτό ή πώς θα γίνει. Και τέλος, θέλω να κάνω ένα παράπονο εδώ, καθώς έχω και λίγο χρόνο. Τις προάλλες ζητήθηκε από αυτή την Επιτροπή Αλίας μία έκθεση ε, που είχε κάνει μία αντιπροσωπεία της DG Mare για την Παππούα Νέα Γουινέα. σε σχέση με το θέμα των πιστοποιητικών ε, αλίας. Ε, ζητήθηκε από αυτή την επιτροπή αυτή η έκθεση και αρνήθηκε η ΓΑΜΑΔΕΛΤΑΜΑΡΕ. ΜΑΡΕ. Για ποιο λόγο και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και είναι τόσο απόρριτο που δεν μπορούμε εμείς οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις ε, μελέτες. Νομίζω ότι είναι η ελάχιστη ενημέρωση που μπορούμε να απαιτήσουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σας ακούω κάθε φορά και θέλω να σας πω το πρώτο που μου έρχεται κατά νου είναι γιατί τόση βιασύνη όταν προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά γιατί ε, θέλουμε ε, να πετύχουμε τους στόχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι και δεν είναι όλοι συνεκτικοί συναφείς μεταξύ τους ε, και δίνεται πολύ έμφαση σε ορισμένες πτυχές, όμως δεν επικεντρωνόμαστε σε όλους. Όταν μιλάμε, το χάρη για την ικανότητα, για το 80%, όταν γίνονται κάποιες δηλώσεις από την πλευρά της Επιτρόπου σε σχέση με το ποιες είναι αυτές οι μελέτες. Ε, κοιτάξτε, εμείς ε, είμαστε ε, εισηγητές, αλλά ούτε καν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάποια έγγραφα για να ξέρουμε τι λένε οι εκθέσεις αυτές. Ε, και μιλώ ως Ισπανίδα και ως Σοσιαλίστρια την Ισπανία την ανησυχεί να υπάρχουν τόσες εκθέσεις. Ε, και ας ε, μην ε, φτάσουμε καν στο θέμα της ραστεχνικής ελίας γιατί δεν υπάρχει καν ορισμός και μένα με ανησυχεί πάρα πολύ όταν μιλάμε για την Μεσόγειο και θέλω να σας ρωτήσω εσύ φτάσατε σε κάποια συμφωνία με την Τουρκία ή με το Ισραήλ γιατί και αυτή είναι στη Μεσόγειο υπάρχει μόνο μία συμφωνία που θα υποχρεώσει όσους αποτελούμε μέρος Τη ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και έτσι θα κατακαιρματίσουμε τη Μεσόγειο και θα πληρώσουν το κόστος μίας ε, λανθασμένης πιθανότητα πολιτικής, ε, τα κράτη-μέλη και δεν θα ληφθούν υπόψη ούτε οικονομικές επιπτώσεις, ούτε οι πολιτιστικές επιπτώσεις, ούτε θα ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση ε, της μικρής και παρακτές ελίας. Δηλαδή εδώ θέλετε να πάρετε μια κατάλληλη απόφαση ή θέλετε απλώς να πάρετε μια απόφαση για να βελτιώσετε την κοινή ελία. Και... Ε, μπορώ να σας πω ότι γενικά συμφωνούμε με τους στόχους, όμως για όσα μας αφορούν και μας στείλουν, τι μέτρα θα πάρετε και για τον προπολογισμό, πώς εσείς θα δαπανίσετε για αυτόν τον τομέα της Ελίας που έχει τόσες πολλές ανάγκες. Ευχαριστώ κύριο Σπυρίλο. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε. Συμφωνώ ε, μέσω απάντηση επίτροπος της συντονιστριά μου για το θέμα της ε, Μεσογείου. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν ήδη θετικές απαντήσεις και είμαι ικανοποιημένο. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τις απορρίψεις Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα σημείο αφετηρίας ε, και πρέπει να κινηθούμε σταδιακά σε αυτό το θέμα. Μια τελευταία ερώτηση. Έρχεται στο νου μου, επειδή τις προάλλες ε, κυρώσαμε στο Κοινοβούλιο την επιτάχυνση σε σχέση με τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την αλία, για τις χώρες που είναι σε καθυστέρηση. Μάλιστα δώσαμε 10% επιπλέον ε, για να αποφύγουμε οι χώρες που έχουν δυσκολία να ε, ενεργοποιήσουν ε, το ιδιωτικό ε, κονδύλι να βοηθηθούν και νομίζω ότι ο μηχανισμός που εντοπίσαμε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χώρες μέσω μιας ισχυρής παρακολούθησης από την πλευρά της Κομισιόν και της Επιτρόπου για να αποφύγουμε το εξής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία να μην ε, καταλήξει όπως ε, κατέληξε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη θαλάσσια πολιτική και την αλία. Δηλαδή θέλουμε να μην έχουμε επικαλύψεις, αλλά θέλουμε μία λύση συνέχειας. Γιατί αν έχουμε επικαλύψη δεν θα καταλήξουμε στους επιθυμητούς στόχους. Ευχαριστώ κύριε Πυρίλο. Κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Επιτροπός αναφέρθηκε στην δυνατότητα να αυξηθούν μέτρα χρηματοδότηση μέτρα στήριξης ε, στη μικρή αλία, στην παράκτη αλία, στην αριστεχνική αλία. Ξέρουμε βέβαια ότι κάθε ελευτική πολιτική πρέπει να οστιάζεται σε ένα μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίω έχοντα κατά νου την εφαρμογή του βασικού κανονισμού το επόμενο έτο, αν εγκριθεί και στο ότι θα τεθούν σε εφαρμογή οι μεταρρυθμίσεις. Η ίδια κυβέρνηση στην Αλία θα έπρεπε να υιοθετεί κάποιες αρχές καλύτερης διαχείρισης για να αριθμιστεί η αριστεχνική Αλία. Και με ποια μορφή και συμφωνώντας με κάποιους συναδέλφους που, που τοποθετήκαν πριν, με ποιο τρόπο η Κομισιόν θα μπορούσε να δώσει κάποια κίνητρα και να προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, δεδομένη της σημασία, αλλά δεδομένου και του ότι λείπουν κάποιοι βιολογικοί, οικολογικοί, κοινωνικοί κοινωνικοί, οικονομικοί δείκτες σε σχέση με την μικρή αλία όπως αποκαλείται και καταλαβαίνετε πως η ανησυχία προκαλείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί και υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με τον ορισμό της αεραστατεχνικής αλίας όπως γνωρίζετε, αλλά καθώς αύριο θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα η Περιφερειακή Επιτροπή, ή να ακούσουμε την Περιφερειακή Επιτροπή που έχει εργαστεί για αυτό το θέμα, εσείς Πώς ε, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις προκλήσεις που τίθεται για τη χρηματοδότηση, τον ορισμό κτλ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Για το πρόβλημα, ή μάλλον ας πω καλύτερα την δυνατότητα που ανέφερε ο κ. Βαλένσα, την δυνατότητα δηλαδή να γίνουν μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης πολλαπλών ειδών. Γιατί μίλησε για την υπεραλίευση της παπαλίνας στην Βαλτική και επειδή είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα στο γάδο φέτος. Θα σας απαντήσω ότι φτιάχνουμε το πρώτο σχέδιο πολλαπλών ειδών για τη Βαλτική θάλασσα, για την αλία στην οποία αναφερθήκατε δηλαδή. Ελπίζω ότι το σχέδιο αυτό θα είναι έτοιμο μέσα στο 2013. Πρόκειται για νέα προσέγγιση, διότι είναι προσέγγιση για το σύνολο οικοσύστημα Χρειαζόμαστε χρόνο διότι χρειαζόμαστε νέα γνωμοδότηση, νέες γνωμοδοτήσεις από την ISIS και θα είναι ένα νέο εργαλείο το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Βαλτική για την αλληλεία αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Μέχρι τότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αν θεωρείτε ότι χρειάζονται, ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε. Αυτό συνέβαινε σε άλλη ε, περιοχή στα ύδατα της Σκοτίας όπου έχουμε τροποποιήσει λίγο τα σχέδια αυτή τη στιγμή βελτιώθηκε το απόθεμα. Πάντως ο καλύτερος τρόπος είναι όντως να γίνει σχεδιασμός για πολλά είδη. Ελπίζω ότι ε, του χρόνου λοιπόν θα έχουμε αυτόν τον πρώτο σχεδιασμό για τα πολλαπλά είδη για τη Βαλτική. κυρία Φράγκα ρώτησε σχετικά με το Μαρόκο. Εγώ έστειλα επιστολή στον ε, Μαροκινό Υπουργό για να τον ενημερώσω με πλήρη τρόπο σχετικά με την εντολή που έχω λάβει από το Συμβούλιο μετά από τις συζητήσεις για το πώς θα συζητήσουμε. Ελπίζω ότι μέχρι τέλους Μαΐου, ίσως και μέχρι τέλους Ιουνίου μπορούμε ε, να έχουμε κάποια νέα. Κάποια νέα θα έχουμε λοιπόν και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε και το Ευρωκοινοβούλιο. Ακόμα θα θέλαμε, ναι, ναι, θα, θέλαμε νέα συμφωνία, το κατανοείτε αυτό, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε βέβαια και τις ανησυχίες της άλλης πλευράς. Σε ό,τι αφορά την υπερβάλλουσα χωρητικότητα, χρειάζεται να βρούμε νέους τρόπους για να οριστεί ξεκάθαρα τι σημαίνει overcapacity, η προβάλλουσα χωρητικότητα. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, εμεί θα είχαμε έρθει εδώ να σας δούμε. Στο μεταξύ θα ρίξουμε το ιδιαίτερο βάρος σε αυτά τα νούμερα των υποδυνάμεων, των ισχύων των κινητήρων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ισχύ κινητήρων και θα δούμε τι στοιχεία μπορούν να μας δώσουν συγκεκριμένα οι χώρες μέλη. Ποτέ δεν είπαμε εγώ τουλάχιστον δεν το είπα, εγώ τουλάχιστον δεν το είπα, δεν ξέρω, ότι έχουμε στην Μεσόγειο 80% υπερχωρητικότητα. Ίσως να μην κατανοήσετε καλά. Αυτό που είπα είναι ότι έχουμε 80% των ειδών που υπεραλλιεύονται στην Μεσόγειο. Αυτό είναι αληθές και είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για την υπόθεση αυτή, για την Παππούα Νέα Γουινέα, τη συμφωνία δηλαδή με την χώρα αυτή και οι πληροφορίε που έχω σχετικά σας ενημερώνω κυρία Φράγκα, δεν γνωρίζω την υπόθεση στην οποία αναφερθήκατε. Γενικά τηρούμε τους ίδιους κανόνες για τις συμφωνίες. Θυμάστε όταν ήσασταν πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας όταν είχαμε συζητήσει αυτά. Εάν υπάρχει κάτι που μπορούμε να δώσουμε, βεβαίως θα ε, σας το υποβάλλουμε. Θέλω το Κοινοβούλιο να είναι απολύτως ενημερό. Θα ε, ελέγξω και θα επανέλθω. Για την δυνατότητα να υπογραφούν συμφωνίες με Τουρκία και Ισραήλ επισκέφθηκα την Τουρκία, ήδη έχουμε μια συμφωνία, έχουμε και ε, συνεργασία, θα έρθουν να μας δουν και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κοινέ επιθεωρήσεις για να βρούμε κάποιες λύσεις. Με το Ισραήλ συζητούμε τώρα την δυνατότητα <clears throat> να συναυθεί συμφωνία για προϊόντα αλίας και με τις άλλες μεσογειακές χώρες επίσης συνεργαζόμαστε, αλλά φαντάζεστε ότι θα χρειαστεί χρόνος Κατανοούμε λοιπόν τα προβλήματα. Νομίζω ότι η GFCM είναι ο σωστός οργανισμός στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. GFCM και ICAT βέβαια. Για το Ταμείο Αλίας και τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κύριος Πυρίλο. Το Ταμείο Αλίας είναι Ταμείο Αλίας και Θαλάσσης. Επομένως δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αλληλεία και στις παράκτιες κοινότητες. Δίνουμε δηλαδή χρήματα για οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της αλίας. Για παράδειγμα, έγιναν πολλές προτάσεις και από εσά και από άλλους ευρωβουλευτές, αλλά και από κυβερνήσεις για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για να δώσουμε να χρηματοδοτήσεις για μεταποιητικές βιομηχανίες, ώστε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αλλιευόμενα ψάρια. Αυτά σκεφτόμαστε τώρα για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω χρηματοδότηση για μεταποίηση. Επίσης για το μαγείρεμα των ψαριών, καθώς και για τον αλλιευτικό τουρισμό ως μέρος του θαλάσσιου τουρισμού. Αν θέλουμε στην περίοδο γονιμοποίησης να μείνουν οι ψαράδες έξω από τις θάλασσες, χρειάζεται να τους δώσουμε κάποιες, κάποια κίνητρα να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Να εξασφαλίσουν κάποιο πρόσθετο εισόδημα. Να, ας πούμε, να καθαρίσουν τις θάλασσες από τα πλαστικά, να μαγειρεύουν τα ψάρια, να τα μεταπιούν. Αυτά κάνουμε λοιπόν. Τα χρήματα πάντως πάνε στους ψαράδες και στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ας το πω έτσι. Τώρα, για τις για τα σκάφη μικράς κλίμακας αλίας. Δεν ε, αναζητούμε νέο ορισμό, διότι δεν έχουμε τέτοιο χρόνο. Ο ορισμός μας παραμένει ω έχει στις προτάσεις μας, διότι τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή το μήκο του σκάφους και η ποιότητα του αλλιευτικού εξοπλισμού είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Αν έχουμε περισσότερους παράγοντες, δεν θα μπορούμε να τους ελέγξουμε. Εσείς βέβαια θα κρίνετε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ολοκληρώθηκε ο διαρθρωμένος διάλογος. Σας ευχαριστώ όλους. Όπως ε, συνήθως ε, θα έχουμε και την αντίστοιχη επιστολή. Θα σταλεί σε όλες τις πολιτικές ομάδες και στη συνέχεια θα σταλεί στη διάσκεψη των Προέδρων. Με τα αποτελέσματα του διαλόγου αυτού σας. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Δεν είναι στην αίθουσα αυτή, είναι σε άλλη αίθουσα η συνεδρίαση στις 9 το πρωί. Στις 10, στις 10, στις 9 είναι η συνεδρία των συντονιστών. Σας ευχαριστώ.